Allez, on va commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ξεκινάμε με την ε, υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Έχει προσθεθεί στην αρχή της συνεδριάσεως ένα θέμα για να μπορέσουμε ε, να έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ε, ανθρωπιστική κρίση η οποία πλήττει το κέρας της Αφρικής. Έχετε άλλες παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο της ημερησίας διατάξεως. Τότε ε, υιοθετούμε την ε, ημερήσια διάταξη με αυτή την αλλαγή. Κύριε Μπέργμαν, Θέλετε να σχολιάσετε κάτι, αν όχι, ε, έχετε λάβει την, ε, ε, τα πρακτικά της 14ης και 15ης Ιουνίου. Αν έχετε παρατηρήσει παρακαλώ να τις επισημάνετε στη γραμματεία μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως, διότι διαφορετικά θα υιοθετηθεί. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν τρέχουν αρκετά γρήγορα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έχουμε μια ερώτηση προς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ευτυχώς δεν έχουμε λάβει τέτοιες ερωτήσεις οπότε θα τους αφήσουμε ακόμη ένα λεπτό για να ανέβουν. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις δεν έχω σχόλια αλλά η κυρία Θεοχάρους έχει να μας κάνει μια ανακοίνωση. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μπορείτε να ξεκινήσετε. Thank you, Madam Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό το οποίο θέλω να θέσω ίσως δεν συνδέεται στενά με τις αρμοδιωτές μας, αλλά θα ήθελα να σας πω δύο-τρία λόγια για την τραγωδία που χτύπησε τη χώρα μου χθες. Χθες εξεράγησαν κάποια εκρηκτικά σε 98 περιέκτες το οποίο είχαν κατασχεθεί πριν από δύο χρόνια από ένα ρωσικό πλοίο. Προχώρησαν από το Ιράκ μέσω Συρίας. Πρόκειται για εκτέλεση οδηγίας ε, του ΟΗΕ, Γαλλία ε, Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρωπαϊκής Ένωση και των ΙΠΑ. Χθε, επίσης είχαμε μια διασωπεργαγιά η οποία έφτασε σε αυτή την αυτική βάση στο νότιο τη ε, Κύπρου, οπότε και είχαμε αυτή την ε, έκρηξη των κοντέινες που έρχαν αυτά τα πάρα πολύ ευαίσθητα εκρηκτικά. Πάρα πολύ μεγάλη αυτή η έκρηξη, της οποίας ε, οι διαστάσεις λέγεται ότι είναι στο 1 τέταρτο της βόμβας της Χειροσύμα. Μίλια μακριά γίνεται το και ήταν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν υπάρχει πια αυτή η ναυτική βάση και ο βασικός σταθμός ε, ηλεκτροπαραγωγής σχεδόν καταστράφει. 70 γενναίοι επί δύο ώρες προσπάθησαν να ζήσουν τη φωτιά, να ακοινώσουν την περιοχή από τους ε, πολίτες. 15 ε, είναι ναυτικοί, τέλο πάντων το πλήρωμα της βάσης, διοικητής, αξιωματική. Έχουμε 62 βαριά τραυματισμένους. Ε, οπότε μιλούμε ότι μετά το πόλεμο του 1984, αυτή η πιο μεγάλη καταστροφή μα έχει πλήξει. Το δε πρόβλημα μα είναι ότι τώρα έχουμε πρόβλημα με την ηλεκτρική ενέργεια, ε, blackouts, ε, διακοπή ηλεκτρικού, δεν υπάρχει πόσιμο νερό γιατί όπως ξέρετε εξαρτώμεθα για την αφαλάτωση μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι απαιτείται ότι είμαστε πάρα πολύ βάλλοντοι, οπότε Χρειαζόμαστε την ελληνική ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε σας παρακαλώ να μας υποστηρίξετε με κάθε δυνατή προσπάθεια όλα αυτά τα οποία προσδοκούμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να μας ανακουφίσει από αυτή την τραγωδία. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. On me dit de préciser qu'on n'a pas d'interprétation. Ε, ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχουμε διερμηνία προς τα Σουηδικά. Ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα θα περάσουμε στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Έχει κάποιες ανακοινώσεις η Κομισιόν. Ε, η Κομισιόν δεν έχει ανακοινώσει για σήμερα. Ευχαριστώ. Σε σχεδόν κάθε συνεδρίαση η Κομισιόν δεν έχει ανακοινώσεις. Θα ήθελα να γίνει μια μικρή προσπάθεια τουλάχιστον να μας παρουσιάσετε τις ε, ανακοινώσεις σας, ε, έστω και με λίγα λόγια, γιατί πάντα είναι δυσάρεστο για μας το ότι δεν μας κοινοποιείτε τις ανακοινώσεις. Θα μπορούσατε τουλάχιστον να ξεκινήσετε να κάνετε αυτό από το φθινόπωρο. Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε για την ανθρωπιστική κατάσταση στο κέρας της Αφρικής. Η ανθρωπιστική κατάσταση μας οδήγησε στο να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη για να συζητήσουμε αυτή την κατάσταση. Η ξηρασία στην περιοχή έχει προκαλέσει μίζωνα διατροφική κρίση, επισητιστική κρίση. Πάνω από 12 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν στην Αιθιοπία, στη Σομαλία και στην Κένια. Για αυτή τη συζήτηση έχουμε την ευχαρίστηση να έχουμε μαζί μας, συγγνώμη για την προφορά μου στο όνομα. Είναι δύσκολο τον κύριο Βίτερμπροντ. Ε, τμήματάρχης ε, του B3, τον κύριο Τζέμο Λοντεζάνη, διευθυντή του γραφείου του Παγκόσμιου ε, Επιστημιστικού Προγράμματος Βρυξέλλες, τον κύριο Τίνταρ Βάλτ, σύμβουλο για τα ανθρωπιστικά ζητήματα στην Oxfam και τον κύριο Βιμ Όλτοφ της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ. Θα δώσουμε στον καθένα το λόγο για μια μικρή ομιλία που δεν θα υπερβεί τα 8 λεπτά. Σας ζητώ να την τηρήσετε. Χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στους χρόνους που δίνουμε στους ομιλητές. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Βίτερμπροντ. Έχετε το λόγο. Well, thank you, Madam Chairman. Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σε Βίτεμπρο την η σωστή προφορά στα Ολλανδικά. Ευχαριστώ πολύ που δίνετε το λόγο στην Κομισιόν. Είναι η κατάλληλη στιγμή που εγείρουμε το ζήτημα της ξηρασίας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στο κέρας της Αφρικής. Έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου αποτελεί την σοβαρότερη, ε, ε, ε, το σοβαρότερο επιστηστικό πρόβλημα στον κόσμο σήμερα. Χθε είχαμε μια ενημέρωση στη Νέα Υόρκη μετά από μια επίσκεψη στο κέρας της Αφρικής και μιλάμε για μια κατάσταση ε, πείνας στις ορισμένες περιοχές Πρόκειται για μια κατάσταση επίγουσα ανάγκη. Το 2011 η φετινή χρονιά είναι από τις πιο ξηρέ χρονιές στη κέρα τη Αφρική ε, τα τελευταία 20 χρόνια. Όπως φαίνεται η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί πριν από τις αρχές του 2012. Για δύο συνεχείς ε, ε, χρόνια. πλέον δεν υπάρχει, σεζόν δεν υπάρχει πλέον βροχή σε περιοχές της Αιθιοπίας, της Ομαλίας και της Κένια και της Κένιας ε, οι άνθρωποι πλέον δεν μπορούν να ε, αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα της ξηρασίας. Ε, αυτή η ανομβρία είχε ως αποτέλεσμα την ελλειπή παραγωγή καλλιεργιών. Η γεωργία έχει σταματήσει. Η κτηνοτροφία από την οποία εξαρτώνται αυτές οι περιοχές ε, έχει εξαλειφθεί, υπάρχει πολύ ψηλή θνησιμότητα των ζώων, αυξημένη πίεση, ε, ελλειπή σπόρη, νερό και οι τιμές των τροφίμων έχουν φτάσει σε υψηρά κόρος. Αποτέλεσμα, εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ε, ανάγκες διαβίωσής τους τα προβλήματα διατροφής σε παιδιά 2-5 ε, ετών ε, έχουν διαδοθεί σε όλη την περιοχή. Οι άνθρωποι βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους, δεν μπορούν πια να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ό,τι έχουν, ό,τι υπάρχει ως μέσο διαβίωσης έχει εξαντληθεί. Πολλοί άνθρωποι απλά επιβιώνουν με ελάχιστα. μιλάμε για 10, 11 ή 12 εκατομμύρια ανθρώπους ε, οι οποίοι υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Στην περίπτωση της Αιθιοπίας, χώρα με τεράστιες δυνατότητες και εκεί 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι σήμερα ε, που εξαρτώνταν από την επισητιστική βοήθεια σήμερα έχουν, αυξηθεί, έχουν φτάσει τους στα 4,5 εκατομμύρια. Ε, αδυνατούν ε, να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ε, ξηρασίας. Δυστυχώς αυτή η επίγουσα επισητιστική κατάσταση θα συνεχιστεί μέσα στους επόμενους μήνες. Εδώ μιλάμε για τις περιόδους κατά τις οποίες οι άνθρωποι χρειάζεται να αντλήσουν από τα αποθέματα, τα οποία ωστόσο είναι ανύπαρκτα, διότι ε, δεν υπήρξε ε, θερισμός. Οπότε βασίζονται απολύτως στην ε, βοήθεια. Λόγω λοιπόν της ξηρασίας και των σωρευτικών παραγόντων των υψηλών τιμών, της θνησιμότητας των ζώων και η πίεση όσον αφορά τους σπόρους δημιούργησε ένα πρόβλημα επιστημιστικής ασφάλειας, ένα από τα σοβαρότερα στον κόσμο. Ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι η πιο σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση παγκοσμίω. Και συναντώντα χθε τον Επίτροπο για να προετοιμάσουμε την αποστολή στο Κέρα την επόμενη εβδομάδα, μου είπε ότι η τρέχουσα κατάσταση στο Κέρα είναι το Πακιστάν του 2011, η η e αιτή των αρχών του 2010. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση. Το χειρότερο και αυτό που ουσιαστικά κάνει την κατάσταση καταστροφική και εξαιρετικά ευαίσθητα, ευαίσθητη, η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των διαφορών διενέξεων στην περιοχή. Έχουμε μετατοπισμένους πληθυσμούς στη Σομαλία, στην Αιθιοπία και σε λιγότερο βαθμό σε κάποιες άλλες χώρες. Αλλά επίσης υπάρχει και έλλειψη ε, χρηστής διακυβέρνησης, ε, ανεπαρκής ε, βιώσιμη ανάπτυξη το κέρας της Αφρικής ε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ε, έχει και πάρα πολλούς μετατοπισμένους πληθυσμούς. Υπάρχουν σχεδόν 750.000 πρόσφυγες από τη, Σομαλία, από τη Σομαλία στο κέρας. Ε, στην Κένια υπάρχει το μεγαλύτερο στρατόπεδο μεταναστών σε ολόκληρον ε, τον κόσμο. Υπάρχουν χιλιάδες μεταναστές εκεί και αναμένεται ότι θα φτάσουν σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία 500.000 ε, οι μετανάστες. Στην ίδια τη Σομαλία έχουμε ένα 1,5 εκατομμύριο μετατοπισμένους πληθυσμούς. Μιλάμε για ανθρώπους εν κινήσει λόγω των διενέξεων στη Σομαλία, αλλά όλο και περισσότερο τώρα λόγω της ξερασίας και των οικονομικών συνθήκων. Οι άνθρωποι αναζητούν βοήθεια και κατάλημα. Στην Αιθιοπία αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός μεταναστών από τη Σομαλία. Σήμερα μιλάμε για 1.700 ε, μετανάστες την ημέρα. Στην Κένια Μιλάμε για 1.300 μετανάστες ε, ε, Σομαλούς την ημέρα. Μιλάμε για 90.000 δηλαδή μετανάστες το μήνα, οι οποίοι μεταναστεύουν, φεύγουν από τη Σομαλία λόγω της έλλειψης ασφάλειας, της ξηρασίας, της επισητιστικής, ε, του επισητιστικού προβλήματος. Όπως καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους. Αυτό επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι δυνατότητες που έχουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να προσφέρουν υποστήριξη είναι περιορισμένες. Στην Ερυθρέα, ε, ένα κομμάτι του κέρατος, η πρόσβαση είναι αδύνατη Έχω ενημερώσει ξανά στο παρελθόν αυτή την Επιτροπή. Η κυβέρνηση της Ερυθρέας δεν διευκολύνει την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και ως αποτέλεσμα αποφασίσαμε να σταματήσουμε τις δραστηριότητες μας εκεί. Είναι αδύνατο να δουλέψει κανείς στην ε, Ερυθρέα. Την κατάσταση στη Σομαλία τη γνωρίζουμε, λόγω της έλλειψης ασφάλειας εκεί δεν μπορούμε να έχουμε ε, πρόσβαση ακόμη και στην Αιθιοπία παρεμβαίνει η κυβέρνηση. Όπου λοιπόν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική αρρωγή λόγω της ξηρασίας, ε, λόγω των διενέξεων, λόγω των μετατοπισμένων πληθυσμών και των επισητιστικών προβλημάτων, ως διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζουμε περιορισμούς ε, στην πρόσβαση. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή τη στιγμή να χτυπήσουμε το κόδωνα του κινδύνου να ευαισθητοποιήσουμε τη διεθνή κοινότητα και να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας. Θα τελειώσω λέγοντας τι κάνει η ίδια η Κομισιόν. Φέτος ε, παρήχαμε 64 εκατομμύρια αυξήσαμε το ποσό σε 95 εκατομμύρια. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε χάρη σε αυτό το ποσό βιώσιμη στήριξη. Εάν δεν φτάσει θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό επίγουσας βοήθειας του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για πρόσθετη χρηματοδότηση. Η Κομισιόν κατανοεί την κατάσταση ε, μετά από τις αποστολές που έγιναν. Ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο τώρα στους ε, ετούντες. Ε, ο κύριος ε, Μπερτσάνη καταρχήν υπεύθυνο του Γραφείου Επισητιστικής Βοηθείας της Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Το προσόν είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να επαναλάβω ε, την, τις ουσιαστικές αρχές τις οποίες ήδη διεκήρυξε ο προλαλής σας διότι ουσιαστικά έχουμε τρία τμήματα του κέρατος της Αφρικής όπου υπάρχει μια πολύ κρίσιμη κατάσταση λόγω των χαμηλών βροχοπτώσεων η Ανατολική Κένια, η Νότια Σομαλία και ε, η ε, νότια πλευρά της ε, Αιθιοπίας. Στις άλλες περιοχές υπάρχουν αυξήσεις τιμών, αλλά εδώ θέλω να σας δώσω ορισμένους, ορισμένα στοιχεία σε αριθμούς, διότι εδώ, επειδή μιλάμε για για βοσκοτόπους και ε, για γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυτές είναι οι περιοχές ε, όπου οι άνθρωποι θα πληγούν περισσότερο διότι ε, το, η απόδοση των δημητριακών πριν από ένα χρόνο δεν μπορεί τώρα να συγκριθεί ούτε κατά ένα τέταρτο με τη σημερινά επίπεδο ακόμη και αν υπάρχει ανταλλαγή προϊόντων ε, ε, πέρυσι ε, όσον αφορά τα δημητριακά βλέπουμε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί ε, σημαντικά από 300 ε, στα 440 μεταξύ ε, πέρυσι και φέτος και για το τεφ που είναι η βασική τροφή στην Αιθιοπία και υπάρχει μία αύξηση των τιμών στις βασικές πρώτες ύλες. Στην Αερόμπη παραδείγματος χάρη η τιμή του αραβοσίτου ήταν τον Ιούνιο, δηλαδή τώρα 450 δολάρια τον τόνο έναντι 370 δολαρίων εις την εχμή των τιμών το Απρίλιο του 2008. Το ίδιο βλέπουμε για τα καύσιμα και ε, όλες οι αγορές θα πληγούν. Εμείς ε, μέχρι εχθές είχαμε μία αξιολόγηση των ατόμων που έχουν πληγεί. Ε, επρόκειτο για 9,8 εκατομμύρια άτομα αλλά Αυτά είναι τα αποτελέσματα πολλών ε, ε, διοργανικών ε, αξιολογήσεων, αλλά υπήρξαν δύο αξιολογήσεις οι οποίες έγιναν το Μάιο και συμπληρώθηκαν τέλος Μαΐου σε δύο βασικές χώρες του κέρατος της Αφρικής, την Κένια και την Αιθιοπία και αυτές οι αξιολογήσεις αποκαλύφθησαν εχθές. Δηλαδή εχθές ο Υπουργός Γεωργίας της Αιθιοπίας δημόσια παρουσίασε την, τις αναθεωρημένες ανάγκες ε, της Αιθιοπίας σε ε, έγγραφα και για την Αιθιοπία αυξήθηκαν από 3,2 εκατομμύρια σε 4,5 εκατομμύρια και για την Κένια από 2,4 ε, στα 3,2 εκατομμύρια. Ε, έχετε τα στοιχεία αυτά με ασκερίσκους που δείχνουν τις αλλαγές αυτές και τώρα ε, φτάνουμε σχεδόν στα 12 εκατομμύρια άτομα τα οποία πλήττονται από αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά την σύγκριση η οποία αναφέρθηκε, η σύγκριση με τα πρόσφατα στοιχεία αλλά ακόμη και αν πάτε πίσω στην δραματική πείνα εις την Αιθιοπία το 84-85 αντιμετωπίζουμε τώρα μία από τις φοβερότερες ξηρασίες στο κέρας της Αφρικής και ε, χρειάζεται προφανώς μία επίγουσα αντιμετώπιση και βοήθεια. Αυτό που θέλω τώρα να σας πω είναι να σας ε, υποδείξω δείκτες της ε, ε, ε, ασιτίας και έχουν γίνει από διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τη UNICEF αλλά και από εμά. Ξεκινάμε λοιπόν με μία μέτρηση όπου λαμβάνουμε σαν σημείο κινήσεως του ΓΑΜ 15% και βλέπουμε 24% στην ε, Αιθιοπία 22% μέχρι 37% στις ε, πιο σοβαρά ε, πληγμένες περιοχές στην Κένια και προφανώς το θέμα αυτό πλήττει ιδίως τα παιδιά διότι ε, αν τέλος Μαΐου, Ιουνίου είχαμε παιδιά τα οποία ε, έφταναν εις ε, το στρατόπεδο Αλαντόντ με 45% ο ποσοστό ασυτείας ενώ θεωρούμε ότι στο 2% χτυπάει το καμπανάκι κινδύνου τα προηγούμενα στοιχεία ήδη παρουσιάσανε, αλλά τεχνικά υπάρχει κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Εμείς μιλήσαμε για 1,5 εκατομμύρια ατόμων που πλήττονται στη Σομαλία αλλά και στην Ερυθρέα και στην Κένια. Ουσιαστικά όμως ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται στην περιοχή θα αυξηθεί διότι οι άνθρωποι δεν έχουν πολλές επιλογές ή θα συγκεντρωθούν σε ορισμένα σημεία όπου θα μπορούν να εντοπιστούν ή θα περάσουν τα σύνορα υπάρχουν διαμάχες βέβαια και σειράξεις και δεν είναι εύκολο πολλές φορές να περάσουν τα σύνορα. Οπότε όπως ε, σας δείχνουμε ε, στην επόμενη διαφάνεια αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τον Ιούνιο καλύπτουμε δια των διαφόρων προγραμμάτων 7,3 εκατομμύρια άτομα σε όλες τις χώρες οι οποίες ε, αναφέρονται στη διαφάνεια αυτή και πρόκειται για επεμβάσεις οι οποίες είτε αυξάνουν την γενική ε, διανομή τροφίμων ή ε, στηρίζουν και επαυξάνουν τα προγράμματα ε, βοηθείας προς ορισμένες χώρες ή αυξάνουμε την θεραπευτική σύντηση διότι ε, ξέρετε ότι το σύστημα ε, λειτουργεί καλά. Θέλω ακόμη λίγο χρόνο. Έχουμε ένα πρόβλημα στην Νότιο Σομαλία διότι όπως είπα προηγουμένως πριν από δύο χρόνια ε, η κατάσταση ήταν επίσης πολύ κακή σε σχέση με τη σύγκριση που κάνουμε τώρα αλλά δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί πρόσφυγες οι οποίοι ε, ε, περνούσαν τα σύνορα από την Σομαλία προς την Κένια ενώ τώρα στη Νότιο Σομαλία Υπάρχει η παρουσία ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεις, ε, ε, υπάρχει ε, μία ομάδα εργασίας που πήγε το 2010 αλλά δεν έχει επιστρέψει εκ τότε. Ξέρετε όμως ότι από την προηγούμενη εβδομάδα το ξανασκεφτόμαστε και θεωρούμε ότι είναι θετικό στοιχείο και ε, κατόπιν αυτού ε, θα ξαναξεκινήσουμε τις επιχειρήσεις μας αφού αναθεωρήσουμε την επιτόπου κατάσταση διότι ε, αυτό που λέει το κοινό δεν είναι υποχρεωτικό ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Οι ανάγκες δεν έχουν αναθεωρηθεί και ε, έχουμε ενημερώσει τα στοιχεία ε, από τις αξιολογήσεις αλλά οι ανάγκες βασίζονται ακόμη στο 9,8 μας λείπει 1,5 εκατομμύριο δολάρια μέχρι το Σεπτέμβριο Σεπτέμβριο και το, το κενό αυτό θα αυξηθεί. Εάν λοιπόν αντιδράσουμε τώρα θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα αργότερα και να μειώσουμε και το κόστος των επιχειρήσεων αργότερα οπότε πρέπει να γίνει ε, μία επένδυση και θα ήθελα ε, το Κοινοβούλιο να προωθήσει αυτή την κίνηση. Ευχαριστώ. Ο καθένας ξεπερνά κατά δύο ή τρία λεπτά γι' αυτό και ο τελευταίος ε, ο μιλητής θα την πληρώσει Τώρα λοιπόν δίνω τον λόγο στον κύριο Τσίνταρ Βόλταρ, ο οποίος ε, συνεργάζεται με την Oxfam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τις μελέτες της Oxfam, η οποία είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που εργάζεται ανά τον κόσμο για να μειώσει ε, τα δεινά, αντιδρά στις κρίσης διατροφής και ε, όπως ε, είπε ο συνάδελφος θα δείτε ότι στο τέλος ε, υπάρχει μία κοινή έκκληση στην οποία συμμετέχει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αλλά και η Oxfam και εάν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος οι αριθμοί θα αυξηθούν. Υπάρχουν δύο ε, ε, εποχές όπου υπάρχουν βροχοπτώσεις αλλά ε, μέχρι το φθινόπωρο δεν προβλέπονται βροχές και μπορεί οι επιπτώσεις να επεκταθούν και μέχρι τις αρχές του 2012 και οι συνάδελφοί μου έχουν επισημάνει τις ελλείψεις τροφίμων και όπου υποσυτίζονται υπερβολικά μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού που υποστηρίζονται κατά 50% σε σχέση με το, το κανονικό επίπεδο. Σε ορισμένες λοιπόν περιοχές δεν είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν βοηθείας. Η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι αφού οι βροχές θα έρθουν ή δεν θα έρθουν σε σε τρεις εβδομάδες θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ε, μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ξηρασία αυτή και σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να παρουσιάσουμε τη βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε ορισμένα άτομα τα οποία είναι συγκεντρωμένα σε στρατόπεδα στην ε, Κένια όπου προσέρχονται κάθε εβδομάδα περισσότεροι πρόσφυγες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ως το δυνατόν περισσότερα άτομα. Βλέπουμε ότι 53% στην Κένια και 43% στην Σομαλία και περιμένουμε ακόμη τους αριθμούς για την Ισουθιοπία χρειάζονται βοήθεια. Σε όλες αυτές τις ε, χώρες πρέπει να δοθεί βοήθεια πριν να είναι πολύ αργά πια. Το πρόβλημα πολλές φορές είναι ότι η προσοχή της διεθνούς κοινώσεως αργεί πολύ ε, να ε, εκδηλωθεί και ε, τα δεν επιλύουμε τα προβλήματα που καθιστούν τα άτομα αυτά ευάλωτα καταρχήν. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα σωστό σύστημα διανομής των τροφίμων και μια διατροφική αλυσίδα. Αυτό οδηγεί στους ανθρώπους να μετακινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει με το να επενδύσει στους μικρούς παραγωγούς, να πατάξει την διαφθορά και αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάθονται στο γραφείο τους σε κάποια χώρα και κερδίζουν χρήματα εις βάρος αυτών των πληθυσμών και είναι δυστυχές αυτό. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και ε, να βοηθούν και ω προς την αλλαγή του κλίματος και επίσης χρειάζεται να αναλυθεί δράση για τις ε, εκπομπές του διοξιδίου, ανεβαίνει συνέχεια η θερμοκρασία και όλα αλλάζουν, επομένως ε, πρόκειται να υποφέρει πάρα πολύ η Αφρική, να στερηθεί 20% μείωση των βασικών ειδών γεωργία παραγωγής Οπότε η μία κρίση έρχεται μετά την άλλη και επομένως ε, αυτή η περιοχή της Αφρικής χωρίς διάλειμμα πλήσεται από τη μία κρίση μετά την άλλη και επομένως θα πρέπει να χτυπήσουμε το πρόβλημα στις ρίζες του. Κύριος ε, Όλτοφ τώρα από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά πιο μακρόπνοα, όχι μόνο τη σημερινή κρίση. Γιατί έχουμε μία χρόνια έλλειψη των διατροφής εκεί. Είναι χρόνιο το πρόβλημα. Γιατί ακόμα και τις χρονιές που δεν έχουμε ξηρασία ε, υπάρχει έλλειψη ειδών διατροφής ανασφάλεια, όπω λέγεται, διατροφική. Έχουμε εδώ κάποια στοιχεία, τα οποία όπως αναφέρουν, στην περιοχή αυτή. Το πρόβλημα χρονίζει και δεν σημαίνει καμία πρόοδος όσον αφορά κάποιε καλύτερες επιδόσεις, είναι κάποια εξαίρεση η Αιθιοπία, αλλά πάντως οι τεθέντες στόχοι για την αντιμετώπιση της πείνας δεν φαίνεται να μπορούν να επιτευχθούν. Το γύρο τη Αφρικής επίσης είναι ένας τόπος με πάρα πολύ μεγάλες ε, προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Πρόκειται για μια περιοχή όπου η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι βασικές απασχολήσεις. Δεν υπάρχουν ελεκτικέ. Γεωργία και κτηνοτροφία έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Πρόβλημα υπάρχει και με την θέση σε εμπορία των προϊόντων. Ε, το περιβάλλον επίσης πλήσεται από όλες αυτές τις ξηρασίες που αναφέρθηκαν. Έχουμε και πλημμύρες από καιρούς καιρών και η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη δεν βοηθάει βέβαια καθόλου. Ο πληθυσμός αυξάνεται Οπότε και αυξάνεται η πίεση εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Γι' αυτό λέμε για μεγάλη ανασφάλεια, προβλήματα προσβασιμότητας και διακυβέρνησης. Σε αυτά τα πλαίσια. Για να δούμε. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την μακροπρόθεσμη ασφάλεια παροχής ειδών διατροφής είναι βασικό σημείο της αντιξέχης μα συνεργασίας. Μιλούμε για α, ε, πολύ σημαντική προσπάθεια σε στοιχεία. Θα το δούμε σε λίγο. Οπότε θα πρέπει να προφροντίσουμε την παραγωγή και την ε, προσβασιμότητα για να αγοραστούν τα τρόφιμα και στο παρελθόν μας είχαν ορθά επικοινωνία δεν προσέχαμε πάρα πολύ αυτές τις πτυχές αλλά και το θέμα της σταθερότητας ε, που έχει να κάνει και με την προπαρασκευή για μελλοντικές κρίσεις. Έχουμε κάποια αισθήματα πληροφορίας όσον αφορά τις κρίσεις και την έλλειψη των διατροφής. Σε αυτό έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ε, οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΦΑΟ και άλλων διεθνών οργανισμών. Οπότε και κατά τον τρόπο να ανακοφίσουμε την περιοχή, να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια και να υπάρχει κάποια μακρόπνοη προοπτική στήριξη. Αν αναφέρεστε όλα αυτά τα στοιχεία, θα φτάσετε στο μισό δις ευρώ για τις τρεις χειρικές χώρες. για πενταετία έως επταετία. Το δέκατο πρόγραμμα αυτό θα καλύψει ό,τι προγράμματα έχουμε, ό,τι μέσα πολιτικής έχουμε και το αυτόματο αυτόματοποιημένο ή αυτόματο πρόβλημα ασφάλειας διατροφής. Για να δούμε τώρα τρία παραδείγματα των προγραμμάτων που έχουμε ξεκινήσει στην Αιθιοπία. PSNP λέγεται στα ελληνικά. Δίκτυα ασφαλείας παραγωγής τροφίμων. Εκεί συμμετέχουν ε, όλοι οι διεθνείς μας εταίροι και εκεί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια τροφίμων και προσπαθούμε επίσης να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι θυγόμενοι για να τους καλύψουμε. Δίκτυα ασφαλείας. Και δεν μιλούμε μόνο για κρίσεις, αλλά και στις άλλες περιόδους όπως πέρσι μιλούμε ότι καλύφθησαν 7,5 εκατομμύρια προσώπων. τι διάφορες ευάλωτε το κοινωνίας όπως ηλικιωμένοι, όρφανα παιδιά. Επίσης προσπαθούμε να βοηθήσουμε και όσον αφορά ε, την προστασία του εδάφους, ε, κοινωνικές υπηρεσίες, δρόμοι, πόσιμο νερό. Επομένω, ε, το πρόγραμμα αυτό από ό,τι φάνηκε βοήθησε πάρα πολύ και για τη, τα ιδιατροφής, πρόσβασιμότητα στη, σε παιδεία, υγεία όμως το πρόβλημα ήταν το να βγει κανείς ή ο κίνδυνος να βγει κανείς από αυτό το πρόγραμμα, από αυτό το δίκτυο ασφαλείας, γι' αυτό και εμείς λέμε ε, ότι είναι κάτι πολύτιμο και από πλευράς μας ενθαρρύνουμε αυτά τα 25 εκατομμύρια τα οποία έχουν καλύψει Βέβαια δεν καλύπτεται όλη η χώρα. Έχουμε τομεί τη υπαίθρου που δεν καλύπτονται. Στην Σομαλία, α πούμε, εκεί που θα βοηθήσουμε όσον την κτηνοτροφία. Στην ε, βορειοανατολική πλευρά της χώρας, εκεί που θα βοηθήσουμε όσον αφορά τις εξαγωγές ζώων, να υπάρχει εκτινοτροφική κάλυψη η επιμέλεια υγειονομική, πιστοποίηση, υποδομές για την κτηνοτροφία. Θα καλύψουμε 105 εκατομμύρια προσώπων σε αυτό το σημείο της χώρας. Και είναι τώρα. Εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης υπαίθρου που έχει δύο πυλώνες. Πρώτα-πρώτα παραγωγικότητα για την γεωργία και εκεί που καλύπτεται ένα ευρύφασμα τομέων αλλά επίσης προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσον αφορά τις, περι... τις ξηρές περιοχές ή τις ημί ξηρές εκεί δηλαδή που υπάρχουν ε, και εθνικοί φορείς για την μετώπιση της ξηρασίας. Ασφάλεια και ασφάλιση για την κτηνοτροφία, για τα ζώα και επίσης ε, προστασία, επιμέλεια των βοσκοτόπων. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ακριβώς αυτή η προσπάθεια πρόνοιας για τις ε, ε, περίοδους ξηρασίας και αναπτυξιακή βοήθεια. Όσον αφορά αυτήν την ε, πολιτική ασφάλειας τροφίμων που την ξεκινήσαμε πέρσι ε, για το κείμενο που επίσης θα ψηφίσετε αύριο προσπαθούμε και στα πλαίσια του αυτομάτου προγράμματος που κάνει την περιοδο 2011-2013 πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο. Πρόσφατα είχαμε από ΕΚΟ και ΝΤΕΒΚΟ μια κοινή ομάδα Task Force για ανθρωπιστική βοήθεια, ανάπτυξη, ασφάλεια τροφίμων. και κάποια διαδικασία διαφορετικών φάσεων. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε και στα δύο μέτωπα, και στο ανθρωπιστικό και στο αναπτυξιακό. εκπαιδεύουμε το προσωπικό και επιτόπου προσπαθώντας να μην έχουμε ούτε επικαλύψεις ούτε κενά στις δράσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στα μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Μπερμάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ζήτημα είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι απλά μια καταστροφή λόγω ξηρασίας ή είναι η αποτυχία μια σειράς πολιτικών. Και εγώ πιστεύω ότι είναι το δεύτερο. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι φυσικά η συνέπεια της αλλαγής του κλίματος σε ξηρές περιοχές όπου οι ξηρασίες είναι πιο συχνές και όπου όταν βρέχει βρέχει άφθονα αλλά η βροχή δεν παραμένει στο έδαφος. Αυτό όμως μας κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι οι πολιτικές προς αυτούς τους αγροτικούς πληθυσμούς είναι ανεπαρκείς. Αυτό οφείλεται σε κυβερνήσεις οι οποίες ε, παραμελούν αυτούς τους ε, ανθρώπους τους ε, κοιτούν περιφρονητικά από τις πρωτεύουσε στο Ναϊρόμπι, στην Αντισαμπέμπα και σε άλλες πρωτεύουσε. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν καλύτερες και να είχαν βοηθήσει να αποφευχθούν τα δράματα που βλέπουμε σήμερα. Επισκέφθηκα την ε, Βόρεια Κένια, την περιοχή Τουρκάνα, ε, πριν από μερικές εβδομάδες με τους συναδέλφους μου και αυτό που είδα μου προκάλεσε σοκ. Οικογένειες που έσκαβαν σε αποξηραμένα ποτάμια για να βρουν νερό. Έσκαβαν με τα χέρια τους. δεν είχαν αγελάδες πια διότι ήταν ε, υπερβολικά ξηρό το περιβάλλον. Μόνο κατσίκες μπορούσαν να ζήσουν σε μια τέτοια περιοχή ε, ως αποτέλεσμα της ε, αλλαγής του κλίματος. Αυτοί όμως οι πληθυσμοί ζούσαν πολύ καλά, είναι ικανοί να ζήσουν σε αυτές τις περιοχές. Εφόσον υπάρχουν ε, υλοποιημένες επαρκείς πολιτικές. Έχουν πρόσβαση σε νερό το οποίο υπάρχει κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Έχουν, αν είχαν πρόσβαση σε ενέργεια, σε υπηρεσίες υγείας, σε εκπαίδευση, σε μεταφορές, σε υπεδομές και όπως ε, μίλησαν, είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές ε, μέσω της μετάδοσης γνώσεων για την κτηνοτροφία. Αυτοί οι πληθυσμοί συμβάλλουν σε μεγάλο κομμάτι του αγροτικού εισοδήματος αυτών των χωρών, παρότι δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που χρειάζονται είναι η δυνατότητα, η άδεια του να διέρχονται από τα σύνορα. Χρειάζονται τη επίλυση των διενέξεων μεταξύ των ε, φυλών ε, που πολεμούν για τους ισχνούς πόρους στην περιοχή. Ορισμένες φορές ε, αυτές οι διενέξεις λαμβάνουν χώρα εδώ και πολλούς αιώνες και δεν μπορούν εύκολα να σταματήσουν. Ωστόσο αυτοί οι πληθυσμοί έχουν μέλλον. Δεν χρειαζόμαστε μόνο επίγουσα βοήθεια. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Όλτοφ να μιλάει για την ανάγκη συσχετισμού της ανθρωπιστικής ε, ε, πολιτικής. Ε. Χρειαζόμαστε περισσότερα από αυτό το ανθρωπιστικό πλαίσιο. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε τις αναπτυξιακές πολιτικές μας σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τις πρέπει να αλλάξουμε τις αναπτυξιακές πολιτικές και όχι τον ανθρωπιστικό τομέα. Οι κλιματικές αλλαγές ε, δεν προκλήθηκαν από αυτούς τους αγρότες. Η αγροτική ανάπτυξη παραμελήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερο. Και χαίρομαι που βλέπω ε, μια σαφώς ορατή ε, μεταβολή αυτής της τάσης από το 2008 και η επισητιστική ασφάλεια θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές μέσα στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Έχω ορισμένε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για την έλλειψη χρημάτων. Ο, τι χρηματοδότηση προσφέρουν τα κράτη-μέλη, τι προσφέρουν ουσιαστικά, όχι δεσμεύονται ότι θα διαθέσουν. Επίσης, ε, επειδή δεν άκουσα ακριβώς τι είπατε για το ποσό που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας παρακαλώ να το επαναλάβετε. Στην ε, Ερυθρέα δεν μπορεί να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε πώς πλησιάζετε τους ανθρώπους. Υπάρχει τρόπος να τους πλησιάσετε εκεί και να τους χρηματοδοτήσετε. Αναφέρατε επίσης ότι πέραν αυτών που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θετικών βημάτων για την ε, διατροφική ασφάλεια, ε, αυτό οδήγησε σε μία βελτίωση των τιμών ή μπορέσατε να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρξουν περισσότερα άτομα τα οποία ε, θα, δεν θα πλήττονται από την κρίση. Επιτύχατε κάτι με το πρόγραμμα. Αν όχι, πέστε μας γιατί. Ε, διότι αντιλαμβάνουμε ότι είναι δύσκολο να βρείτε τους ανθρώπους αυτούς. Είναι όμως ο μόνος ρόγος Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν καλυφθεί οι άνθρωποι από αυτό το πρόγραμμα. Και τέλος ε, υπάρχει και μία πιο λεπτομερής ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρηματοδοτεί την εξαγωγή ε, των ζώων. Πού, προς τα πού όμως πρόκειται για περιφερειακές εξαγωγές. Και θα πρέπει να Υπάρχει διασύνδεση μεταξύ της βραχυπρόθεσμης βοήθειας με την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και θα πρέπει να υπάρξει μία πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση διότι πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να μπορέσει κανείς να ξεκινήσει προγράμματα που θα σας οδηγήσουν ε, στο στόχο τον οποίων επιζητείτε. Έχουν γίνει ορισμένες πρόοδοι αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι μία μακροπρόθεσμη θεσμοί πρόκληση όπου θα πρέπει ε, όλοι να φροντίσουμε να παρακολουθούμε όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Θεοχάρους. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπέρμαν ότι αυτό που συμβαίνει στο κέρας της Αφρικής είναι μια σειρά αποτυχιών, σειράς πολιτικών συν την κυβερνητική διαφθορά που είναι πάντοτε παρούσα και την κακή διακυβέρνηση. Θα ήθελα να σας πω ότι όταν έγινε ο μεγάλος λοιμός του 83-84 τον οποίο αναφέρθηκε ένας εκ των ομιλητών εμείς ως φοιτητές στη Θεσσαλονίκη είχαμε αλωνίσει την πόλη και είχαμε συλλέξει μια τεράστια ποσότητα τροφίμων και χρημάτων για να τα αποστείλουμε στην Αιθιοπία και να σας θυμίσω βέβαια όσοι μπορεί να θυμάστε αυτό το γεγονός την ίδια μέρα τα αεροπλάνα της Αιθιοπίας βομβάρδιζαν την Ασμάρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την συγκυρία που νομίζω ότι είναι τραγική και δείχνει ότι δεν έχουμε πλέον συνέστηση του ποιε είναι οι πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Από τη μια να ξεποδαριαζόμαστε για να μαζέψουμε βοήθεια και από την άλλη να ακούμε ότι βομβαρδίζουν ένα γειτονικό λαό. Σε αυτή την υπόθεση τρεις παράγοντες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρώτον, οι διεθνείς οργανισμοί και χαίρομαι που ακούσαμε την συνεισφορά τους, οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται με την διανομή τροφίμων και σε αυτό το θέμα νομίζω ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια με τα συμπληρώματα διατροφής, με το γάλα σε σκόνη που μπορεί να σώσει πάρα πολλά παιδιά και με την καλή διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών. Με συγχωρείτε. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι πληθυσμοί της Αφρικής αυτοί καθεαυτοί, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν και να γίνεται προσπάθεια στις μικρές κοινότητες. Και αυτό αναφέρθηκε και συμφωνώ απόλυτα. Έχω την εμπειρία εδώ και 16 χρόνια να δουλεύω με μικρές κοινότητες στην Αφρική, να παρακάμπτουμε την κυβερνητική διαφθορά και να βλέπουμε ότι οι κοινότητες αυτές ποτέ δεν στερούνται ούτε το ΜΕΙΣ, ούτε έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια από το εξωτερικό. Ευτυχώς αυτές, αυτά τα προγράμματα αντιγράφονται σε μερικές περιπτώσεις είτε από τοπικές κυβερνήσεις είτε από τοπικές αυτοδιοικήσεις και γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη των ε, επαρχιών των μεγάλων χωρών που μαστίζονται από την πείνα. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ εδώ είναι η χρησιμοποίηση της παραγωγής για βιοκαύσιμα. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο απιά τους α, αφρικανικούς λαούς, αλλά τους στερούσε το φαγητό. Δηλαδή όταν η παραγωγή του καλαμποκιού διοχετευόταν μαζικά για την παραγωγή βιοκαυσίμων, καταλαβαίνετε ότι δεν έμενε κάτι για να μετατρέψουν σε μέις και να, και να τρώνε. Ε, δεν ξέρω αν αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. Πάντως στις νότιες περιοχές της Αφρικής προσπαθήσαμε και νομίζω το έχουμε ε, ελέγξει. Και ο τρίτος παραγοντάς είναι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί από τους οποίους ξεκινάει η βοήθεια προς την Αφρική. Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη υποφέρουμε από hyperalimentation, από υπερκατανάλωση τροφίμων, από κατασπατάληση των τροφίμων και είναι απαραίτητο να υπάρξει μια επανεκπαίδευση του ευρωπαϊκού πληθυσμού ούτω ώστε ούτε να γίνεται αυτή η υπερκατανάλωση και ό,τι διασώζεται να μπορεί να αποστέλλεται σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, και ήθελα και εγώ να παρέμβω, οπότε συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε η κυρία Θεοχάρους και ο κύριος Μπέρμαν σήμερα το πρωί. Χρειάζεται πολιτικό θάρρος και πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι του, η έλλειψη του πολιτικού θάρρους ε, εκ μέρους όλων, για να πούμε την αλήθεια έχει φτάσει η ώρα να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά και την κερδοσκοπία που ανέφερε ο κύριος Βάη της Oxfam διότι διαβάζω πολλά επ' αυτού και έχει φτάσει η ώρα ε, ε, υπάρχει πληροφόρηση στην Ευρώπη και στην Αμερική ε, για υπερκατανάλωση στις πλούσιες χώρες αλλά εάν δεν πατάξουμε την κερδοσκοπία και τη διαφθορά διαφθορά δεν θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να επιλύσουμε το πρόβλημα. Είναι θέμα πολιτικό. Όλες οι πολιτικές ε, ομάδες, όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να ξεπεράσουν ε, αυτό το σκεπτικό και γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλους τους εκλεγμένους, σε όλους τους βουλευτές να έχουμε το θάρρος να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να πατάξουμε την κερδοσκοπία γιατί είναι ντροπή. Δεν μπορούμε πλέον να τα δεχθούμε αυτά σήμερα τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κόρτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Αλλά πρώτα πρώτα σας ευχαριστώ για το έργο σας, για αυτό το πρόγραμμα για την ε, διατροφή ε, της Oxfam ε, όλων των μη κυβερνητικών όλων των διεθνών φορέων για τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όπως ε, είπαμε θα ε, είμαι σύντομο, διότι πιστεύω ότι έχει ξεκαθαριστεί το πόσο είμαστε ενωμένοι όσον αφορά την δέσμευσή μας για την ε, αντιμετωπίσουμε την πείνα αλλά και την κλιματική αλλαγή και προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια και η Ευρώπη και ο υπόλοιπο κόσμος και εάν όμω δεν κάνουμε κάτι το αποφασιστικό για την αλλαγή του κλίματο δεν θα πιάσει τόπο καμία προσπάθεια. Η κατάσταση του γέρος Αφρικής είναι μια κατάσταση που κάθε τόσο επιδεινώνεται, υποσχεώζει τα ίδια προβλήματα και προσπαθείτε εσείς, προσπαθεί όλη την κοινότητα, όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί, να προσπαθήσει και με οικονομική συμβολή, ακριβώς όπως έκανε στο Πακιστάν για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ θλιβερό το να έχουμε 12 εκατομμύρια τα οποία να βασανίζονται εκεί και να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πάντως και πάλι συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείται, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκεί επί τόπου ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε τι γίνεται. Τον Αύγουστο θα τα πούμε που θα πάω στην Αιθιοπία και θα αποκτήσω άμεση εποπτεία του τι γίνεται. Μπορείτε να υπολογίζετε στην αμέριστη συμπαράστασή μας. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις εκτός από κάποιες ε, λεπτομέρειες που θέλω να ε, ρωτήσω για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν ερωτήσεις. Εν συντομία, κυρία Πρόεδρε, ε, για κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις ήθελα. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ολοκληρώσω αυτά που υπάρχει αρχικά. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 98 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής ε, για τις χώρες του κέρατος οι συμβολές ε, το 2011 όλων των κρατών μελών είναι 83 εκατομμύρια αν το συγκρίνουμε με τις ανάγκες ε, των υπολείπων οργανισμών να αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα. Είναι ένα σημαντικό ποσό, αλλά χρειάζεται να κινητοποιήσουμε περισσότερα. Το ζήτημα ε, της Ερυθρέας φυσικά είναι ευαίσθητο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εάν δεν υπάρχουν συνθήκες σωστής εργασίας για τη διεθνή ανθρωπιστική κοινότητα, είναι αδύνατο να εργαστούμε θα πρέπει να αποφύγουμε την κατάχρηση των, των χρηματοδοτήσεών μας. Δεν θέλουμε τα χρήματά μας να καταλήξουν σε στρατιωτικές ομάδες. Δεν έχουμε ελευθερία κινήσεων. Με δυσκολία μπορούμε να πάρουμε μια βίζα. Δεν μπορούμε να φύγουμε από την Ασμάρα. Δεν μπορούμε να προβούμε σε ανεξάρτητη αξιολόγηση των αναγκών. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στους αποδέκτες. Δεν έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες γενικότερα είναι κλειστός ο χώρος για την ανθρωπιστική αρρωγή. Δεν υπάρχει ε, τρόπος να φτάσει η ανθρωπιστική ε, διεθνής κοινότητα στους αποδέκτες ε, και όσο εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτούς, αυτοί προσπαθούν να έρθουν σε εμά. Βλέπουμε πόσοι διέρχονται από τα σύνορα προς την Αιθιοπία και το Σουδάν. Όσον αφορά την επιστημιστική ανασφάλεια, δεν το είπα, αλλά έπρεπε να το είχα πει φυσικά, ότι Σήμερα παρέχουμε μία επίγουσα απόκριση σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Από το 2006 έχουμε δώσει πολλά κονδύλια για ετοιμότητα σε περίπτωση ξηρασίας προσπαθώντας ε, να θωρακίσουμε τις κοινότητες αυτές σε τοπικό επίπεδο οικοδομώντας υποδομές στις τοπικές κοινότητες. Αυτό κάνουμε από το 2006. Μπορώ να σας δώσω αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό έγινε αποτελεσματικά. Υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία από τους εταίρους μας, ε, από την Oxfam και από τους υπόλοιπους, ότι ό,τι κάνουμε προσπαθώντας να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινότητες βοήθησε στο μετριασμό των συνεπειών της ξηρασίας. Ευχαριστώ. Δεν ε, είχα κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τα μέρη του Κοινοβουλίου που εξέρουν το έργο της ανθρωπιστικής κοινότητας. Ήθελα να επανέλθω εν συντομία σε ένα ε, σημείο. Κάθε φορά που έχουμε ανθρωπιστική κρίση αναφέρουμε το γεγονός ότι ότι δεν είχαν γίνει αρκετά αναπτυξιακά έργα, ότι οι κυβερνήσεις δεν ήταν αρκετά υπεύθυνε. Δυστυχώς όταν φτάνουμε στην αιχμή μιας ανθρωπιστικής κρίσης, ε, με συγχωρείτε, ε, όταν, φτάνουμε, όταν αρχίζουμε να ξεπερνάμε σιγά σιγά μια ανθρωπιστική κρίση, τείνουμε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Κάτι που επαναλαμβάνω συχνά αυτή στις μέρες είναι ότι Εάν ε, οι κυβερνήσεις δεν ακολουθούν, ε, δεν παίζουν έναν πολιτικό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ένα τέτοιο ρόλο για την αντιμετώπιση της επισητιστικής ασφάλειας με τον τρόπο που το κάνουμε σήμερα ε, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Δεν είναι ότι τα αποτελέσματα είναι κακά σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και θετικά παραδείγματα κυβερνήσεων που έχουν πραγματική πολιτική βούληση και μέσω πολιτικών διαδικασιών βγάζουν τους ανθρώπους από συνθήκες φτώχειας, από καταστάσεις επισητιστικής ανασφάλειας και υποσυτισμού. Και εδώ μιλάμε κυρίως για τον αγροτικό πληθυσμό, για τους βοσκούς του κέρατος της Αφρικής, αλλά και για άλλε μικρές πληθυσμιακές ομάδες όλο τον κόσμο. Είτε πρόκειται για οικονομική κρίση, είτε για ανθρωπογενή καταστροφή. Οι άνθρωποι δυστυχώς ως αποτέλεσμα πέφτουν σε καταστάσεις οι οποίες απαιτούν ανθρωπιστική επέμβαση. Πρέπει λοιπόν να μιλάμε για όλα αυτά όχι μόνο όταν έχουμε ανθρωπιστική κρίση, πρέπει να ε, θέσουμε ως προτεραιότητα στην ατζέντα την επιστημιστική ασφάλεια υπό, σε όλες τις εποχές, ακόμη και αν δεν υπάρχει κρίση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Συγγνώμη, κύριε. Madam Chair, there three questions. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω τρεις, υπήρχαν τρεις ερωτήσεις σχετικά με τις εξαγωγές κτηνοτροφίας από την Σομαλία. οι, ε, ιδίως ε, οι καμήλες ήταν προς τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη. όσον αφορά την Αιθιοπία και το πρόγραμμα, εάν μπόρεσε να δημιουργηθεί η δυνατότητα να μην περιπίπτει κανείς ε, στη φτώχεια μόλις υπάρχει μία κρίση. Όντως υπάρχει ε, αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή αποφεύγουν οι άνθρωποι να πουλήσουν τα μικρά ζώα τους και είναι πιο εύκολο να επανέλθουν στις ε, τακτικές τους ασχολίες ε, μετά από την πάροδο της ξηρασίας. Ε, προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτές τις δυνατότητες, αλλά συγχρόνως υπάρχει ένας ε, μηχανισμός όταν ε, υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές μπορεί κανείς να διευρύνει το δίκτυο ασφαλείας σε μια ευρύτερη περιοχή και μιλήσαμε ε, για τις ε, γεωργικές δραστηριότητες και τη βοσκή και ιδίω τη βοσκή ε, που δεν επηρεάζεται από το δίκτυο ασφαλείας διότι όταν καταρτίστηκε το 2005 το δίκτυο ασφαλείας ξεκίνησε με τις, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, και μετά προχώρησε στους βοσκοτόπους και αυτό όχι τόσο πολύ στη Σομαλία. Επιπλέον πολλά εξαρτώνται από τα δημόσια έργα και τα δημόσια έργα εξελίσσονται εκεί που οι άνθρωποι ζουν για περισσότερο χρόνο. Οπότε είναι δυνατόν να τους προσεγγίσει κανείς ενώ εάν μετακινούν κινούνται συνέχεια είναι πιο δύσκολο να τους βρούμε. Τελειώνω το λόγο. Όχι. Καλώς. Λέει πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Α, συγγνώμη. Κυρία λόγο. Αναφέρθηκε το τι ευκαιρίες υπάρχουν και νομίζω οι ειδικοί που έχουμε καλέσει μπορούσαν να μας πούν τι πιστεύουν. Από ό,τι κατάλαβα, η βιολογική γεωργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί απαιτώντα λιγότερα εργαλεία και νερό. Και αυτό θα βοηθήσει, ιδίως τους μικροκαλλιεργητές. Συμφωνείτε? ή νομίζετε ότι θα βοηθούσε περισσότερο η νομιζετε οτι θα βοηθουσε περισσοτερο η τεχνολογια Θα σας αφήσω να απαντήσετε. Η ερώτηση είναι πολύ εύστοχη. Το ερώτημα αυτό είναι πιο ευρύ από απλά το κέρας της Αφρικής, από αυτό που μιλάμε, που συζητάμε τώρα. Υπάρχουν διαφορετικές ε, συνθήκες ε, σε κάθε περιοχή του κόσμου, σε κάθε αναπτυσσόμενη χώρα και οι ε, δυνατότητες οι τεχνολογικές δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ανακοίνωση της Κομισιόν ε, περισσυνή σχετικά με την επιστημιστική ασφάλεια. όπου αναφέρεται η, αγροοικολογική εντατικοποίηση. Χρειάζεται να εντατικοποιήσουμε την ε, γεωργική παραγωγή λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά για να επιτευχθεί αυτό, με, αλλά αυτό πρέπει να επιτευχθεί με βιώσιμο τρόπο. Ε, τα παραδείγματα που έχουμε σε αυτό το τομέα μοιάζουν ε, πολύ, πλησιάζουν πολύ τις οικολογικές προσεγγίσεις. Πιστεύω ότι αξίζει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, ενδεχομένως σε κάποια επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, ε, ε, να συζητήσουμε τους διάφορους τύπους ε, γεωργίας, μιλάμε για βιολογικά προϊόντα και για άλλες διαδικασίες. Ίσως πρέπει να το εξετάσουμε με τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο η αποστολή παρατήρησης του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τους εμπειρογνώμονες που ήταν εδώ και που φεύγουν τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για τις παρατηρήσεις σας. Ε, παρουσίαση λοιπόν των συμπερασμάτων της ε, ε, αποστολής ε, παρατήρησης των εκλογών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Σαντσισνέρα είναι καλεσμένος να συμμετέχει σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Δυστυχώς δεν μπόρεσε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, προεδρευόταν από τον κύριο Μπελμπα και δίνω το λόγο αυτή τη στιγμή. Ε, κυρία ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας συνοψίσω το τι ισχύει μια μικρή εισήγηση, τι έγινε σε αυτές τις εκλογές ακριβώς όπως είπατε, τον Απρίλιο του 2011, που πήγε, κλήθη να ψηφίσει ο Λος του Περού για, για, για τις δύο βουλές της χώρας, 50% και ένα. Συν ένας ήταν η, το, το, το, το, το κριτήριο να πέρασαν στο δεύτερο γύρο, τον Ιούνιο επομένω ε, έγινε ο δεύτερος γύρος με τους ε, δύο επικρατέστερους ε, υποψηφίους, ο Μάλα και ο Φουχιμόρα. Οι δύο παρατάξεις τους και κατόπιν της υπουργής των εκλογών πήγαμε εκεί για διάσκεψη των Προέδρων επίσης είπε ότι πρέπει να πάμε εκεί 3 με 6 Ιουνίου του 2011. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου απαρτιζόταν από την κυρία Φεραγούτου, την Εστέρα Θεία και Κάρλος Ιτουργκάης από το ΕΛΚΑ, Ενεργία Γκερέρο, Λουίς Γέγεθ από τους σοσιαλιστές, τον κύριο Μίτσελ Καμίνσκι του ECR και εγώ από την Άλντε ως ε, πρόεδρος. διαπιστώσαμε ότι τρέχει αναπτύξη με 7% το τελευταίο 5%. Υπάρχει σταθεροποίηση τη χώρα Το 2008 ε, φτάσαμε να ανάψει 10% που είναι ρεκόρ για τη χώρα. Παρά όμω αυτή την ανάπτυξη, οι κοινωνικέ συνθήκε είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, κάτι το οποίο διαπιστώσαμε και εκεί με τι επαφέ που κάναμε. Η... Τα στοιχεία σχετικά με την ε, φτώχεια είναι πάρα πολύ ψηλά και μιλάμε για 60 70% σε μερικές των άνδρων που είναι κάτω από το κατόφυλλο της φτώχειας. Ε, τώρα, χαμηλά, ε, 10% του ΕΠ τα, χρήματα τα οποία θα πάνε κυβέρνηση για την κοινωνική πολιτική. Βεβαίως και ενδιαφέρεται έντονα το κοινοβούλιο και το πέρο. Φερόμαστε για την πολιτική κατάσταση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως επίσης και για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τη μετάβαση δημοκρατία. Το 2002 και όπως ξέρετε έχουμε αποφανθεί με ψηφίσματα πάρα πολλές φορές. Επίσης θα πρέπει να σας τονίσω εν κατακλείδη ότι έχουμε μια εμπορική συμφωνία με Κολομβία και Περού. Συνήφθη τον Μάιο 2010, αλλά ακόμα δεν έχει κυρωθεί. Εδώ ε, και στις βουλές των χωρών εκείνων. Στον πρώτο γύρο, όπως είπαμε, κανείς δεν έλαβε αρκετές ψήφους για να είναι αυτόνομη κυβέρνηση. Οπότε η κατανομή των ψήφων στους τρεις αρχικούς υποψηφίους, Σύσκη, Τολέδο και Καστανιέδα, τελικά ο Μάλα με 31% πήρε την πρώτη θέση και Βούχη Μόρι με το Φόρθα 2011 την παράταξή του που πήρε 23,5% των ψήφων. 130 ήταν οι εκλεγέντε στην πρώτη περίοδο και ο περίεργο είναι ότι ο Τολέδο, ο οποίο ήρθε τέταρτος στις προεδρικές, ήταν η τρίτη δύναμη στις κοινοβουλευτικέ. Επίση θα πρέπει να σα τονίσω ότι νόμος του 2000 όριζε το εκλογικό σύστημα και όριζε ότι θα πρέπει να υπάρχουν 30% γυναίκες στα ψηφοδελτία. Οπότε, από 29% το 2006 των γυναικών θα είναι 22% το 2011. Ο Φουχημόρη, η Φουχημόρη είναι η πρώτη γυναίκα που συμμετέχει έτσι στις εκλογές. Αυτό, 750.000 είναι ψήφοι που έπεσαν από το εξωτερικό, που, που έστειλαν. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι υποχρεωτική η ψήφος στη χώρα και από τα άλλα στιγμή μας έδωσαν προκύπτει ότι κάποιοι οι οποίοι έχουν πεθάνει ε, δεν έχουν ληφθεί υπόψη από τα στατιστικά στοιχεία και επίσης πάρα πολλοί προτιμούν να πληρώσουν το πρόστιμο παρά να πάνε να ψηφίζουν. Φυσιολογικά εξελίχθηκαν οι εργασίες μας στα πλαίσια της αποστολής παρατηρητών που είχαμε αναλάβει. 70 ήταν οι από 25 χώρε. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία μεταξύ της αντιπροσωπείας και των κοινοβουλευτικών πήγε πάρα πολύ καλά. Με τον επικεφαλής ε, της εκλογής επιτροπής και με άλλες πρόσωπες της χώρας ήρθαμε σε επαφές, συζητήσαμε διάφορα όπως την προεκλογική εκστρατεία, τον ρόλο των ΜΜΕ, τα εκλογικά προγράμματα, τα διάφορα γκάλο που είχαν γίνει, σχέση με την Ένωση, ήταν τα βασικά σημεία που συζητήσαμε. Είπαμε, είδαμε την Φουχημόρη, τον Ουμάλα, τον Τολέδο, τον, τον κύριο Κοτσίνσκι επίσης. Επίσης, την Εκλογική Επιτροπή και το, ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους του Βουλίου Εξωτερικών Επίση στη Λίμα ήταν όλοι οι πρέσβει των χώρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Οργανισμού των Άνδεων. Επίσης, εν παραδείγματι, βλέπετε και μία σύνοψη των εκδηλώσεων που κάναμε. Ήμασταν πάντως κατά την ψήφιση, κατά το κλείσιμο των καλπών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας επίσης. Πήγαμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών για να δούμε πώς ερχόντουσαν από το εξωτερικό οι ψήφοι των εκπατρισμένων και πώς λαμβανόντουσαν υπόψη την καταμέτρηση. Είναι όπως έπρεπε. Πήγαμε επίσης και στα γραφεία της μη κυβερνικής οργάνωσης που λέγεται Διαφάνεια Πάρα πολύ θετικό είναι ο ρόλο τη μη κυβερνητική αυτή οργάνωση. 5.000 ε, ήταν εκείνοι που για αυτόν τον μη κυβερνητικό οργανισμό ε, καθόντουσαν και βλέπαν ε, ανά τη χώρα τι καταγγελίες υπήρχαν. Είχαμε 20 εκατομμύρια ψηφοφόρους και είχαμε 300 ενστάσεις πέσα από τις οποίες εξετάστηκαν την ίδια μέρα των εκλογών. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ήταν οριακά τα αποτελέσματα, ήταν ε, τις πιο δύσκολες εκλογές για τα κόμματα, η ε, ε, πόλωση υπήρχε, αλλά... Όπως έλεγα προηγουμένως, αυτό οφείλεται στην έντονη αντιπαράθεση των δύο βασικών υποψηφίων και αυτοί που τα είχαν, έλεγαν τα 40% δεν θα ψήφιζε τον Ουμάλα με τίποτα και το 39% έλεγε ότι ποτέ θα ψήφιζε τη Φουχημόρη. Είναι αυτοί όμως που πέρασαν το δεύτερο γύρο. Η Φουχιμόρη είχε ελαφρά ε, περισσότερος, περισσότερη προτίμηση και φαινόταν θα κερδίσει. Όμως, από όλες μας επαφές πρόκειψε ότι αντιστράφει τα τελευταίες μέρες και το βλέπουμε αυτό. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Επειδή βάστον σου στην προβλητική εκστρατεία, τέλος πάντων, η ομάδα έκανε κάπως συναισθηματικά φορτισμένη προεκλογική εκστρατεία. Και θεωρήθηκε ότι είναι πιο εθνικιστική η πλατφόρμα. Η ΔΕ Φουχημόρ ήταν πιο, όχι πιο λαϊκιστική, αλλά λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένη ε, εκστρατεία. Προεκλογική επίση. Εντυπωσίασε το ότι ο πατέρας της υποψήφιας, ο Βούχη είχε κάνει πολλά για τους ε, ηθαγενείς της χώρας. Αυτό αναδείχθηκε πάρα πολύ. Το προέβαλε Φουχημόρη πάρα πολύ. Αλλά υπήρξαν πάρα πολλοί δυσάρεστοι χαρακτηρισμοί και πολύ και οφείλεται ακριβώς σε αυτήν την παράθεση η αλλαγή, η αντιστροφή της τάση που υπήρχε στι προτιμήσει του λαού. Επίσης, αβεβαιότητα. Υπήρχε τα τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών. Η Φωγημόνη μα είπε ότι εάν κερδίσει ο αντίπαλος θα τον συγχαρεί όπως και έκανε Στη δε συνέντευξη τύπου τονίσαμε πέντε σημεία. Πρώτα-πρώτα που ήταν σωστή η εκλογική διαδικασία και η καταμέτρηση. ηλεκτρονική ψήφος που έγινε σωστά. Η συμμετοχή των γυναικών. Η προσβασιμότητα που είχαν οι ανάπηροι να ψηφίσουν. Ο ρόλος των ΜΜΕ που παρακολουθήσαμε πάρα πολύ στενά και εν συμπερασμένη θα πρέπει να πούμε ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και σε δύο μήνες θα υποβληθούν οι συστάσεις μας προς την κυβέρνηση της χώρας. Η αποστολή μας ήταν να παρακολουθήσουμε τις εκλογές στο Περού αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό το οποίο επισημάνω μπορούν να εφαρμοστούν σε πάρα πολλέ χώρε όπω α πούμε η πλαισίωση των ε, αναπήρων και το πώ θα βοηθούν να ψηφίζουν. Αυτό θα μπορούσε να είναι παράδειγμα για τι χώρε τη Ευρώπη, όπω επίση και η ηλεκτρονική ψήφο, που ήταν πολύ πετυχημένη προσπάθεια, θα μπορούσαμε και αυτό να το μεταλαμπαδεύσουμε σε ευρωπαϊκέ εκλογέ και έτσι να είναι εκλογέ πιο διάφανες. Γι' αυτό θα βοηθούσε και την εικόνα των κομμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την αρκετά εκτενή αναφορά. Αν κάποιο από τα μέλη θα ήθελε το λόγο, ο κύριος Κορτές. Ε, θα είμαι πολύ ψήφι. σύντομος. Πρώτα-πρώτα να συγχαρώ την πρόεδρο της ε, Επιτροπής των Παρατηρητών των Εκλογών για άλλη μια φορά θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο και πολύ σημαντικό ο ρόλο του Κοινοβουλίου στην ε, περίπτωση αυτή. Είχα την ευκαιρία να πάω στο Περού. Πήγα πριν από λίγου μήνε στα πλαίσια τη κοινότητα των Άνδεων, είδα την κυρία Φουχημόρη, τον κύριο Ομάλα, και πριν από 6-7 μήνες επίσης είχα κάποιες επαφές ε, κατά τη διάρκεια της προλογική Εκστρατεία. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την Πρόεδρο τι γίνεται, τι έγινε με τον ε, Μάριο Βάργας Λιώσα τον ρόλο του να στηρίξει ε, υποψηφίους και με την αλλαγή της στάσης του την τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ, λέει πρώτος. Α, συγγνώμη. Έχετε το λόγο, ναι. Βιάστηκαν παρά το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια να δώσουμε σε όλους, όλους όσους πήγαν εκεί και στην ε, αποστολή της ε, Ένωσης αλλά και στους ε, τεχνικούς που ήρθαν μαζί μας, σε όλους ε, όσους βοήθησαν όσον αφορά το έργο της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Ο Μάριο Βάργας Λιώσα τώρα και ο Λεχάνδρο Τολέδο. Όχι, τελικά δεν μπορέσαμε να, τον συνα... να τους συναντήσουμε, τον Λιώσα τουλάχιστον, αλλά είναι αλήθεια ότι υπεστήριξε έντονα τον υποψήφιο. Τι να σας πω, δεν έχω τις πληροφορίες. Όσον αφορά τον Αλεχάνδρο Τολέδο, τον είδαμε και αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι στον πρώτο γύρο είχε 33% της προτίμησης του λαού. Έκανε μια κανονική υπολογική εκστρατεία με χαρακτηρισμούς προς ε, τους ε, αντιπάλους του όπως ο κ. Κοντσίνσκι είναι μαθητής μου, μαθητευόμενος διατέλεσε έλεγε. Αυτό δεν εκτιμήθηκε από τον κόσμο αυτή η χαρακτηρισμή και γι' αυτό και δεν εισέπραξε την εκτίμηση του κοινού στην τελική ψήφο. το δεύτερο γύρο. Επομένω θα μπορούσε να περάσει, αλλά τότε που βρεθήκαμε εκεί ήταν φανερό το πόση ένταση υπήρχε γιατί ο κόσμος φοβόταν για το πού πάει η χώρα. Ε, είχαν στο μυαλό τους το τι έκανε ο Τσάβε στη Βενεζουέλα, από την άλλη μεριά υπήρχαν προοπτικέ φιλελεύθερες εξέλιξεις. Και ο ρόλος του, το λέω, ήταν το ότι ακριβώς είχε αναλάβει την ευθύνη του να εξισορροπήσει τις εξελίξεις μετά την νίκη του Μάλα. Εξού και οι επαφές του με οικονομικούς και στο Περού και στις ΗΠΑ που είχε μεταβεί. Και σας είπα τι είναι στον πρώτο γύρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, δύο άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Έχουμε ακόμα τρία λεπτά. Δεν είστε υποχρεωμένοι να πάρετε το λόγο αν δεν θέλετε. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, κ. Βιάρντο. Ε, κυρία Πρόεδρε, ναι. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σύντομα σχόλια. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες των εκλογών. Ε, ήδη μας τις εξήγησαν με μεγάλη σαφήνεια. Υπάρχουν απλά θέλω να πω ορισμένες πτυχές ενδιαφέρουσες ε, που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ως αποστολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μεγάλη προβολή στο Περού κατά τη διάρκεια των εκλογών. Χάρη στην παρουσία της αποστολής παρατηρήσης των εκλογών η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε ε, συχνά στον τοπικό και στο διεθνή τύπου ε, όσον αφορά τις εκλογές ε, στο Περού. Υπήρξε λοιπόν ε, σημαντική προβολή της δράσης της Ένωσης στο Περού και γενικότερα στη Λατινική Αμερική χάρη σε αυτή την αποστολή. Δεύτερο σημαντικό σημείο αυτή η αποστολή παρατηρήσεις των εκλογών μας επέτρεψε να ενισχύσουμε τις πολιτικές μας διμερείς σχέσεις με το Περού. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η η αποστολή είχε πολύ καλές επαφές ε, με τον κύριο Μάλα και αυτό ανοίγει έναν πολύ ικανοποιητικό δρόμο για να συνεχίσουμε να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο με το Περού. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι επιθυμούμε να θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτικό παράγοντα στις σχέσεις μας με το Περού που ενδιαφέρεται σε θέματα διακυβέρνησης, δημοκρατίας και ανάπτυξης και όχι μόνο εμπορίου. Όχι μόνο για τον επιχειρηματικό κόσμο, ε, πολλές φορές ε, αυτό βλέπουμε στις σχέσεις μας με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ενίσχυση λοιπόν των πολιτικών σχέσεων με το Περού. Και επίσης μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Περού και στη Λατινική Αμερική. Ενισχύθηκε χάρη σε αυτή την αποστολή, χάρη στον επαγγελματισμό, την αμεροληψία και το πολιτικό όραμα της αποστολής. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την εικόνα ενός σημαντικού πολιτικού παράγοντα στο Περού και στη Λατινική Αμερική και επίση ε, για να ολοκληρώσω από την άποψη της παρατήρησης των εκλογών υποστήριξη ε, της δημοκρατίας και της διακυβέρνησης πιστεύω ότι αυτή η αποστολή στο Περού μας επέτρεψε να διατηρήσουμε ένα σημαντικό γεωγραφικό ε, ισοζυγίο, μια σημαντική γεωγραφική ισορροπία στην περιοχή ε, διότι πρόκειται για μια περιοχή όπου πρέπει να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και αυτή η αποστολή για το 2011 ήταν η πιο σημαντική αποστολή που είχαμε στη Λατινική Αμερική. Σε γενικέ γραμμές αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Μάλιστα πιστεύω ότι μιλήσαμε για όλα. Ας περάσουμε στο σημείο 6, χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Τον Αυρελίο η Κομισιόν εξέδωσε μια ανακοίνωση για την ενίσχυση της ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη ανάπτυξη εν ώψη τη αξιολόγηση ε, τη ε, δημόσια στήριξη. Αναφέρονται οι πρόοδοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στον τομέα της αναπτυξιακής αρρωγής, ε, επίσης όσον αφορά τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών η Επιτροπή μας ε, προετοιμάζει ένα προφορικό ερώτημα προς την Κομισιόν και, και ένα ψήφισμα για μια από τις επόμενες ολομέλειες. Σήμερα έχουμε καλέσει την Κομισιόν να μας παρουσιάσει την ανακοινωσή της. Έχουμε επίσης καλέσει το ε, CPDM, το ECPDM έχετε στους φακέλους σας τα σχετικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη διαχείριση της αναπτυξιακής πολιτικής. Έχετε το λόγο για το πολύ 10 λεπτά. Θα κάνω την παρουσίαση εν ονόματι της ε, Επιτροπής ε, διότι θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω ε, για την συμμετοχή του Κοινοβουλίου διότι έχουμε ετοιμάσει ορισμένα σχέδια τα οποία και μπορείτε να τα ξεφυλίσετε συνεχίσετε όσο θα μιλάμε. Ε, ο συνάδελφος Ιρασό ε, στα δεξιά μου είναι στη διάθεσή σας να σας απαντήσει αν έχετε ερωτήσεις. Πρέπει να σας πω περτίνος είναι η ε, έκθεση Καταρχήν πρόκειται ε, για τα διάφορα θέματα της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν ε, αναφέρεται στην Επιτροπή ούτε εις την εσωτερική δράση μετά το 2013 δηλαδή στο νέο πλαίσιο. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για τις αποφάσεις οι οποίες οδήγησαν στην απόφαση της Δόχα για την ανάπτυξη το 2008 να παρακολουθούμε την πρόοδο, την επίτευξη των στόχων και να παρουσιάζουμε στο Συμβούλιο μια ετήσια έκθεση το Συμβούλιο παρακολουθεί ότι ε, εφαρμόζουμε τις επιταγές και τώρα επιπλέον υπάρχει μία ε, ε, πλέον αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και την απόδειξη ότι προωθείται όντως η ανάπτυξη των χωρών που ενισχύονται ε, και ε, παρακολουθείται και ε, η κατάσταση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη. Ε, ε, ε, όσον αφορά την πέτηση των πολιτικών αρχηγών το 2010 παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητήθηκε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και νομίζω ότι προχωρήσαμε σε αυτό το θέμα βλέπουμε ότι υπάρχει μία έκθεση που δεν έχει σχέση με τα άλλα θέματα όπως το παρελθόν Υπάρχει μία συνοπτική ε, ε, έκδοση η οποία θα ε, δημοσιευτεί για το κοινό και επιπλέον οι απαντήσει στο ετήσιο ερωτηματολόγιο για να παρακολουθούμε την πρόοδο στην οποία ε, βασίζεται ε, η έκθεσή μας διότι τώρα ε, έχουμε απαντήσεις από όλα τα 27 κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν αναρτηθεί σε μία ιστοσελίδα και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Ποια θέματα καλύπτει το πρόγραμμα. Καταρχήν, τις ε, ε, επόμενες δεσμεύσεις που έχουν σχέση με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε, Ενώσεως και της αναπτυξιακής βοηθείας της. Καταρχήν το θέμα φορολογίας και αναπτύξεως για να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η βοήθεια και πόσο αναπτύσσεται η το εμπόριο και να δούμε ε, πώς προωθείται η συμμετοχή των ε, ε, αναπτυσσομένων χωρών στα διεθνή θεσμικά όργανα. Βλέπετε πόσο διάφορες πηγές υπάρχουν για χρηματοδότηση ε, ιδίως ε, εις ε, τις υποανάπτυξη χώρες αλλά για μας η αναπτυξιακή βοήθεια είναι πιο ο σημαντική πηγή γι' αυτό και πρέπει να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, της ε, ενσωματώσεως του 7% αναπτυξιακής βοηθείας ε, στο πρόγραμμά μας και να έχουμε μία ημερομηνία για την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή το 2015. Εν τω μεταξύ, ήδη το 2002 είχαμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε δύο φάσεις. Καταρχήν, συνδυασμό των ιδιωτικών και δημοσίων στόχων, ε, και μετά να προχωρήσουμε μέχρι το 2015. Συλλογικά υπάρχει ο στόχος του 2006. Υπάρχουν βέβαια χώρες που δεν έχουν πετύχει το στόχο αυτό, αλλά τώρα ε, δεν επιτύχαμε το στόχο αυτό λόγω ενός ε, ελλείμματος 15 δισεκατομμυρίων. Το βλέπετε ή στον πίνακα. Κινητοποιήσαμε λιγότερο από το 56% που επιζητούσαμε και ο στόχος αυτός ε, δεν επέτυχε ε, ε, τους, τις προβλέψεις τις οποίες είχαμε καθορίσει ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις συλλογικέ της ε, ε, δεσμεύσεις για το 2010. Για το 2015 θέλουμε να κινητοποιήσουμε την βοήθεια συλλογικά για το 2015. Ορισμένοι βρίσκονται κάπου παραπάνω και η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει ε, να ε, βοηθήσει επίσης. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να επιτύχουμε τον στόχο και να έχουμε 55 ε, δισεκατομμύρια σαν χρηματοδότηση ε, και αν συνεχιστεί η πορεία που επετεύχθη το 2004 με 2010 θα χρειαστούμε 25 χρόνια ακόμη και όχι 5 χρόνια για να επιτύχουμε τον στόχο του 0,7% πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να λάβουν έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο το οποίο θέλω να τονίσω εδώ, ότι δηλαδή ε, έχουμε δεσμευτεί να υπάρξουν στοιχεία και να υπάρχει μία καλή απόδοση με μείωση ε, των ε, φιλοδοξιών ε, αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αφρική, ε, προς ε, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που επίσης είχαμε, δεν πετύχαμε το στόχο του 2010 αλλά τουλάχιστον σε μικρότερο ποσοστό και ε, οι δωρητές παρουσιάζουν καλές αποδόσεις και μπορείτε να το δείτε από το τελευταίο πίνακα και έχετε και ένα διάγραμμα που δείχνει πώς μεμονωμένα επιτυγχάνονται οι στιόχοι. Ε, όσον αφορά τα κράτη-μέλη ε, θελήσαμε να επιβεβαιώσουμε την συλλογική δέσμευση να ε, υπάρξει μία εθνική προσπάθεια κατά τρόπον ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι, να βελτιωθεί η αποδοτικότητα ε, των μεμονωμένων προγραμμάτων αναπτύξεως για τα επόμενα κράτη και άρα βλέπουμε ότι δεν έχουμε ε, άγνωστους νέους στόχους, είναι οι δεσμεύσεις οι οποίες είχαν αναλυφθεί ήδη από πέρυσι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα χαράς διαπιστώνουμε ε, ότι επιτυγχάνουμε τις δικές μας δεδηλωμένες προθέσεις προς τα, τις χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη ουσιαστικά να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα που είχαν, στα οποία είχαν καταλήξει πέρυσι. Προτείναμε πολλά, αλλά τώρα όλη η ημερήσια διάταξη αναθεωρείται ε, φέτος και για την βοήθεια ε, για το εμπόριο επίσης έχουμε ε, διατυπώσει συγκεκριμένα συγκεκριμένες προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τους ε, νέους μηχανισμούς με δυνατότητα αναγεννήσεως και ε, ε, βλέπετε ή στα συμπεράσματα της ανακοινώσεως που καταλήξαμε. Η έκθεσή μας έγινε ικανοποιητικά αποδεκτή από το Συμβούλιο, αλλά ε, όχι όλοι, ε, όλοι οι στόχοι δεν είχαν επιτευχθεί και δεν καλύπτονται από την έκθεση και επιπλέον ε, είδαμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτησε την ε, έκθεσή μας αλλά θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για να επιτευχθεί ο στόχος μας. Πιστεύουμε ότι χάθηκε μια ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα και σε άλλους τομείς και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα διότι θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς την οικονομική κρίση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν το οποίο διαπιστώνουμε από πλευράς του Κοινοβουλίου είναι κάποια σκέψη για το πόσο το Κοινοβούλιο θα βοηθήσει την ε, Επιτροπή ε, όσον αφορά την ανάπτυξη και θα επανέλθω προς συζήτηση αλλά εφόσον υπάρχει άλλος ομιλητής ο οποίος θα συμπληρώσει θα παραμείνω εδώ. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ διότι όντως εάν όλοι ξεπερνούν το χρόνο τους δεν θα ε, επιτύχουμε. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας, δεν είναι ευχάριστο για μένα, αλλά τώρα τον λόγο έχει ο κύριος ε, Λαπόρτ για 8 λεπτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το ECDPM είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που εξετάζει τις ε, διάφορες σχέσεις. Ε, έχουμε ανεξάρτητους ε, εταίρους για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Θα ήθελα να σημειώσω τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι χαίρομαι που βλέπω ευρύτερη προοπτική πέραν της αρρωγής για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής βοήθειας. Όλοι γνωρίζουμε από εμπειρία ότι τα χρήματα από μόνα τους ε, δεν επιφέρουν ανάπτυξη. Αυτό έχει αναγνωριστεί σε όλες τις σημαντικές δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός. Ακόμη και σε επίπεδο της Αφρικανικής Ένωσης και των Αφρικανικών Οργανισμών που αναγνωρίζουν ανοιχτά ότι εν τέλει η ανάπτυξη αποτελεί ευθύνη των κυβερνήσεων και των πληθυσμών των αναπτυσσόμενων χωρών. Οπότε έτσι έχουμε μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση της ανάπτυξης και δεν εστιαζόμαστε μόνο στις επίσημες αναπτυξιακές αρρωγές της όντα. Όχι μόνο στην ποσότητα της αναπτυξιακής αρρωγής, γιατί υπάρχουν και πολλά περισσότερα που πρέπει να εξετάζουμε. Αυτό ήταν ένα από τα ωφέλη αυτής της ε, έκθεσης ε, υπευθυνότητα. Ε, ήταν η πρώτη φορά που συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κινητοποίηση των τοπικών πόρων, ε, τις ε, ικανότητες, τις επενδύσεις, ε, καινοτόμες χρηματοδοτήσεις, να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, τη συνοχή πολιτικής, επειδή αποτελεί φυσικά ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη θα λάβει χώρα. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν θετικά, θετικές ενδείξεις, μπορούν να συμβάλλουν στην μεταμόρφωση των κοινωνιών. Γνωρίζουμε απόλυτα ότι ε, πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική πρόοδο. Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 500 σελίδες, πολύ υλικό για ανάγνωση για όσους δεν εργάζονται εδώ. Αλλά πιστεύουμε ότι παρέχει μια σωστή αξιολόγηση του όσον αφορά το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις κοινέ μας δεσμεύσεις. Από αυτή την άποψη χαιρόμαστε ιδιαίτερα που πρόκειται για ένα αρκετά άμεσο ανοιχτό έγγραφο που καταδεικνύει τις ε, κοινέ ευθύνε ότι υιοθετεί μια προσέγγιση που προσπαθεί να ε, πάει πιο πέρα από τις επίσημες αναπτυξιακές αρρωγές. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε ότι χρειαζόμαστε καλύτερη διακυβέρνηση, καλύτερα φορολογικά συστήματα ουσιαστικά για την κινητοποίηση των εγχώριων πορών εκτός φυσικά από όλα τις υπόλοιπες, τις υπόλοιπες επενδύσεις που χρειάζεται να γίνουν για να συμβαλούν στην ανάπτυξη. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ καλή διαπίστωση της εκθέσης. Επίσης είναι ιδιαίτερα επικριτική της, εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι οι πολιτικές πρέπει να έχουν συνοχή με τους στόχους. Ε, τονίζεται λοιπόν η συνοχή πολιτικής ε, ως τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει καλύτερες επιδόσεις. Θα μπορούσε να επενδύσει περισσότερο. Ε, ας δούμε ποια είναι οι ελλείψεις αυτής της φιλόδοξης έκθεσης. Υπάρχουν κάποια μικρά κενά όσον αφορά την υλοποίηση. Σε... Θεωρούμε ότι η έκθεση τονίζει υπερβολικά αυτούς τους ODA, αυτούς τους στόχους ODA αυτός ο στόχος δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Ας είμαστε ρεαλιστές. Λέμε συστηματικά ότι μέχρι το 2015, αυτό είναι σε τέσσερα χρόνια από τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εποχές οικονομικής κρίσης θα κινητοποιήσει ή θα ξοδέψει επιπλέον 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακή αερογή μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Είναι ε, παράλογο να λέμε κάτι τέτοιο, ας είμαστε ρεαλιστές. Ε, Έχω λίγο απογοητευτεί επειδή η έκθεση και η παρουσίαση της Κομισιόν δεν εστιάζεται περισσότερο σε άλλα ζητήματα πέραν των ODA. Ε, απογοητεύουμε που δεν έχουμε συζητήσει πέρα από αυτό το ζήτημα του 0,7 που φυσικά είναι σημαντικό αλλά δεν είναι και το μόνο δεν είναι ε, ο μόνος χρηματοδοτικός πόρος που πρέπει να εξετάσουμε θα ήθελα λοιπόν η Ένωση να είναι και πιο φιλόδοξη όταν ε, προσπαθεί να εξετάσει άλλους πόρους ε, χρηματοδότησης πέρα, πέραν των LDA. Μέχρι στιγμής βλέπουμε περιορισμένη γνώση της φορολογικής διακυβέρνησης. Υπάρχουν τα προγράμματα για αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν επίσης πολλά προβλήματα στη συστηματική αξιολόγηση της πολιτικής οικονομίας των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν τη φορολογική τους κινητοποίηση. Έχει νόημα να επενδύσουμε ένα σωρό και να χρησιμοποιήσουμε κοινοβούλια, υπεύθυνου οργανισμούς ή να εγκαταστήσουμε ή να υλοποιήσουμε φόρους όταν γνωρίζουμε ότι το πολιτικό καθεστώς δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά για όλους αυτούς τους πολιτικούς θεσμούς. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη πολιτική ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις διαφορετικές χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υποστηρίξει αυτή τη νέα φορολόγηση και την κινητοποίηση ε, άλλων πόρων. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα. Θα δώσουμε πόρους σε χώρες που δεν κάνουν προσπάθειες ε, να βάλουν λίγα εξετάξει τα χώρια πράγματα. ποιες διαφορετικές προσεγγίσεις πρέπει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες που έχουν ξεφύγει από τη σωστή οδό, πώς θα πρέπει εμείς ως Ευρωπαίοι να γνωρίζουμε καλύτερα τι κάνουμε, ώστε να επιτυχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα βάσει της πολιτικής συνοχής. Βλέπουμε και εδώ μια αντιστροφή της τάσης. θα ήθελα να πω ότι ο συμπεράσμα ότι η λύση δεν είναι περισσότερη αρρωγή αλλά μια νέα προσέγγιση της αναπτυξιακής αρρωγής βάσει της συνυπευθυνότητας των διαφόρων παραγόντων των ε, Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, ε, των οργανισμών ε, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και των ίδιων των αναπτυσσόμενων χωρών και η εφαρμογή της διαφοροποίησης διαφόρων πόρων για τη χρηματοδότηση. Όλα αυτά μαζί μπορούν να έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη. Ποιο θα μπορούσε να είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι έχει παραμεληθεί λίγο σε αυτή την ανακοίνωση της Κομισιόν. Δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, ενώ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Θα μπορούσε να εκδίδει προειδοποιήσεις ε, σε περιπτώσει αντιστροφής τάσεων σε σχέση με τα όσα διακηρύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε ε, ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ε, την τρέχουσα τάση στα περισσότερα κράτη-μέλη της ε, εθνικοποίησης ε, κατά κάποιο τρόπο των αρρωγών όπου το κάθε κράτος μέλος θέλει να αποκομίσει ωφέλη από την αρρωγή που προσφέρει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια κατανομή των εργασιών, να υπάρχουν κοινοί προγραμματισμοί να μην δίνουμε, προσφέρουμε μονομερή αρρωγή από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο τέλος θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι είναι σημαντικό με αυτή την έμονη ιδέα που έχουμε, είναι λίγο άσκημος αυτός ο όρος που λέω, αλλά αυτή η αιμονή που έχουμε να ε, αποκομίσουμε κάτι για τα χρήματα που δίνουμε ε, και αυτό μπορεί να εμποδίσει κατά κάποιο τρόπο τις ε, τις επενδύσεις μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που είναι απαραίτητες και των οποίων τα ωφέλη ίσως να μην είναι απολύτως ορατά άμεσα και που ενδεχομένω αποτε, αποτελούν, χρειάζονται περισσότερο χρόνο ώστε να επιτευχθούν μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση. Κάνω έκκληση λοιπόν προ τα κρατη και στα κοινοβούλια, ώστε να είμαι βέβαιο ότι η μακροπρόθεσμη πτυχή τη ανάπτυξη δεν θα παραμεληθεί προ όφελο μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση που, όπω βλέπουμε, ε, εμφανίζεται σε πολλά κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στου ε, βουλευτέ και πρώτο θα το λόγο ο κύριο Κάσμερικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε και κύριοι, σας ευχαριστούμε για τα όσα μας είπατε. Η αναπτυξιακή βοήθεια ίσως δεν είναι η καλύτερη μορφή που χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε τις ε, αντισόμενες χώρες. Όμως, αποδεικνύουν τη συνέπεια της πολιτικής μας σήμερα. Ήμουν ε, στην συνεδρίαση της ε, Επιτροπής της Γεωργίας, όπου η Προεδρία παρουσιάζει τις προτεραιότητές της. Και ορισμένοι βουλευτές διατύπωσαν κάποιες προτάσεις. Ελέγχθη ότι με αυτές τις προτάσεις θα ήταν δυνατόν να πετύχουμε περισσότεροι συνεπείς πολιτικές μας και άλλες προτάσεις οι οποίες θα έφεραν το αποτέλεσμα όπως ας πούμε κάποιες ε, πολιτικές απορρίθμισης, κάποιο διαχωρισμό ε, των αρμοδιοτήτων των ε, κοινών οργανώσεων αγοράς Μιλούσαν επίσης και για κάποιο παγκόσμιο οργανισμό, ο οποίος θα αναλάμβανε ε, την διαχείριση της ροής των γεωργικών προϊόντων, την θέση του σε εμπορία, την προστασία των αγορών, ε, την αντιμετώπιση των εξαγωγείων κλπ. Όμως, θα πρέπει κάθε πολιτική να διέπεται από συνέχεια. Έχω τώρα δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Με τι ρυθμό αυξάνονται οι δαπάνες, οι για την αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αφρική. Σε κάποια κρατημέλη υπάρχει πραγματικά υποχρηματοδότηση για κάποιες χώρες τουλάχιστον. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Μήπως μπορεί να μας πει η Επιτροπή πώς θα πετύχουμε τη βελτίωση αυτού του 2%. Πώς δηλαδή θα, θα πείσουμε τα κρατη να αυξήσουν την ε, προοικοδότηση. Πώς θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις μας για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται επομένω για έναν κίνδυνο που εδώ ελοχεύει. Γιατί υπάρχουν κάποια κρατημέρια τα οποία δεν συμβάλλουν αρκετά, αλλά ταυτόχρονα μειώνουν την ήδη μικρή τους συμβολή. Όπως και η Πολωνία και άλλες χώρες. Τα λίγα θα τα κάνουν λιγότερα. Τι λέτε, πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό το φαινόμενο. Ο επόμενος. Όσα ελέγχθησαν μου δίνουν κάποιες ε, ιδέες εκτός από τις προκαταρκτικές μου παρατηρήσεις γιατί φυσικά και θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική η βοήθεια και δεν είναι θέμα μόνο ποσοτικό, έχει σημασία ε, για το πώς ε, τρέχει το σύστημα, πώς θα το βελτιώσουμε, πώς θα γίνεται καλύτερη ίσπραξη των φόρων. Όλα αυτά ε, μας απασχολούν. Πρέπει να δούμε τώρα για τα πιο συγκεκριμένα σημεία της βοήθειας. Να έχουμε μόνιμο προβληματισμό όσον αφορά όλους τους εμπλακωμένου, όλες τις κινήσεις που γίνονται. Εγώ όχι, δεν θέλω να ενταχθώ στο 0,7% αλλά υπάρχουν και άλλες μεταβλητές στο, πρόγραμμα, στο πρόβλημα αυτό. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Λαπόρτ, αυτό το οποίο μα εξήγησε, γιατί ακόμα και αν όλα όλα γίνουν τόσο πρέπει να γίνουν, θα χρειαστεί και αυτό το 0,7% επιπλέον ε, σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, η οποία δημιουργεί ανισότητε μέσα στην ίδια τη χώρα, στην δεδομένη χώρα, παρά μεταξύ διαφορετικών χωρών. Πέραν αυτό τώρα. Κάτι για τους δωρητές. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζεται αυτό το επονίδιστο φαινόμενο το οποίο σημαίνει ότι ανεχόμαστε αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Δηλαδή, θα πρέπει κανείς να ρίξει μια ματιά στο σχετικό κατάλογο που έχουμε γιατί έχουμε τρεις-τέσσερις κατηγορίες χωρών, έχουμε εκείνους οι οποίοι είναι πάνω από το 7%, η Δανία, Σουηδία, κάτω χώρε και Λουξεμβούργο. Οι κάτω χώρε απεφάσισαν από το 0,9 να πάνε στο 0,7% οπότε ακόμα και αν καλύπτουν τον τεθέντα στόχο όσον αφορά το σύνολο των 27 και αυτοί, οι Ολλανδοί δηλαδή, συμβάλλουν στην συρρήγνωση των προοπτικών. Και υπάρχουν επίσης κάποιες χώρες, επομένως, που είναι υποδειγματικές, δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι προσεγγίζουν το στόχο ε, σιγά σιγά μέχρι το 2015 να καλύπτουν το στόχο της χρηματοδότησης Ας πούμε Ιρλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, ίσως και άλλοι, που είναι κάποιες χώρες ε, ή υποδειγματικές σε σχέση με αυτό. Και, επομένω, κάνω αυτό το οποίο πρέπει σε σχέση με ό,τι συμφωνήθηκε. Πολύ καλό. Επομένω, υπάρχουν και άλλη μια κατηγορία χωρών οι οποίοι δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο που έχει τεθεί, όπω η Γερμανία. Είναι εκπληκτικό παρά τα, τις ε, οικονομικές τους επιδόσεις. Τρία χρόνια μετά την κρίση σχεδόν έχουν λύσει το πρόβλημα. Και η Ιταλία βέβαια, για γνωστούς λόγους. Ε, οπότε χωλαίνει εκεί πέρα το, το θέμα. Επίσης, υποδειγματική είναι και η Βρετανία. Το νημερό Βασίλειο με όλες τις περικοπές που γίνονται παντού δεν έχει κάνει καμία περικοπή όσον αφορά την αντιστοιχική βοήθεια. Αυτό είναι προς έπαινο. Άρα, πού καταλήγουμε. Ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίε δεν κάνουν τίποτα για να πιάσουν το στόχο παρά το ότι ακμάζουν οικονομικά και άλλες παρά την κρίση την οποία περνάνε τα πάνε πάρα πολύ καλά. Επομένως, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Άρα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα άλλα του κ. Λαπόρτ με βρίσκουν σύμφωνα. Όμως θα πρέπει να επιμείνουμε όσον αφορά αυτό το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό Δηλαδή είναι θέμα πολιτικής καταφέρει κάτι. Ευχαριστώ το λόγο όχι τώρα Ή θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο ή όχι. Γιατί δικαιολογιε υπάρχουν πολλές. καλο ο κακο καιρός είναι θέμα το κανει θέλει να καταφέρει κάτι. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ σχετικά με αυτά που ελέγχθησαν περί πολιτικής βούλιες, γι' αυτό αποτυγχάνουν χώρες σαν τη Γερμανία και άλλες, διότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε το 0,7% σαν στόχο γιατί μόνο εάν δημιουργήσουμε αυτή την τεράστια πίεση θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, αρχηγού, ε, χώρες οι οποίες θα ντραπούν που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους διότι διαφορετικά θα μας πούν ε, δεν μας ενδιαφέρει το ότι δεν επιτυγχάνουμε το στόχο στόχο, δεν μας ενδιαφέρουν ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτές της αποτυχίας και πιστεύω ότι το, ο στόχος του 0,7% είναι πολύ σωστός παρόλο που δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας βοηθήσει και ε, στους αριθμούς που έχουμε τώρα βλέπουμε ότι κρύβονται πολλοί αριθμοί οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται πραγματικά ε, στο, στα ποσά τα οποία καταλήγουν στις υποανάπτυξη χώρες σχετικά με το PECD, την διόρθωση της πολιτικής ανάπτυξης, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά πρέπει να αναφερθεί σε δυσάρεστα θέματα όπως τα βιοκαύσιμα και άλλα που ίσως δεν θέλουμε να κοιτάξουμε ε, και να εξετάσουμε ή θέματα όπως το εμπόριο και τα λοιπά. Επίσης το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και πρέπει να συμβάλλει στην αναπτυξιακή βοήθεια διότι διαφορετικά δεν ενδιαφέρονται οι άλλοι για το ότι γίνεται εδώ και αυτό ίσως ε, είναι κάτι που δεν βλέπουμε τόσο πολύ στην ομάδα μας αλλά ε, πρέπει να υπάρχει εσωτερική συνοχή στο Κοινοβούλιο να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτή την προοπτική. Συμφωνώ ότι υπάρχει μία δυσάρεστη τάση για το value for money, δηλαδή την αποτελεσματικότητα όπου όλοι στο τέλος αυτό που θέλουν να πούνε ναι, οικοδομήσαμε 500 σχολεία χωρίς να αποδείξουν πόσο βελτιώθηκε η παιδεία λόγω αυτού και αυτά συμβαίνουν πριν την συνάντηση στο Μπουζάν όπου πρέπει να αναθεωρήσουμε όλο μας το πρόγραμμα διότι αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότης ε, και αλληλενημέρωση διότι ε, ουσιαστικά σε κάθε σχέση υπάρχουν δύο μέρη είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε. Πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί, να αποφύγουμε να υπάρξει κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά διαπιστώνουμε ότι έχουμε δυσκολίες να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Έχω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα να έχουμε αυτή την ε, έκθεση και επίσης θα φανεί ε, τι όντως ε, αντιμετωπίζεται σοβαρά από τα κράτη-μέλη και πώς υπάρχει κάποια επαφή με τις με τα κοινοβούλια των, αναπλε... υποανάπτυξη χωρών και πόσο παρακολουθείται η εξέλιξη αυτή εκεί. Πρέπει και εμείς να είμαστε υπόλογοι στους πολίτες των υποανάπτυξη χωρών, στους βουλευτές τους και στην κοινωνία των πολιτών τους. Τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Μπέρμαν. Νομίζω ότι η κυρία Κέλλερ μας κάλυψε όλους. Η κυρία Κέλλερ μας κάλυψε όλους, διότι ε, από σεβασμό για την ε, ε, γλώσσα μου θα μιλήσω Ολλανδικά σχετικά με το 0,7%. Μόνο ο, ένας προϋπολογισμός στις πλούσιες ε, χώρες ε, ανατιμάται ε, αυτομάτως σε κάθε χώρα. Είναι ο προϋπολογισμός ανάπτυξης. Αυτός βελτιώνεται εάν η, χώρα, η οικονομία πάει καλά καλά και μειώνεται αν ε, η οικονομία πάει κακά. Δηλαδή αντικατοπτρίζει την κατάσταση της οικονομίας μας. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε ο στόχος του 0,7% αναπτυξιακής βοήθειας να το σεβαστούμε διότι επηρεάζει την δικιά μας ευημερία ακόμη και αν κοστίζει παραπάνω 500 ε, δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βρουν άλλους ε, πόρους και άλλα έσοδα για να μπορέσουν να ε, σεβαστούν αυτό το στόχο. Παραδείγματο χάρη η φορολόγηση των συναλλαγών μπορεί να ενισχύσει τα κράτη-μέλη και να τους προσφέρει μία επίσημη ε, προσθήκη στην αναπτυξιακή βοήθεια και ε, ε, επίσης για ορισμένα μέτρα που πρέπει να αναλυφθούν στο θέμα το κλιματολογικό. Δεν πρέπει δηλαδή να απογοητευτούμε και να λέμε ότι δεν θα επιτύχουμε το στόχο αυτό και συμφωνώ ότι ε, θα πρέπει αυτό το θέμα να, πρέπει να το ξαναεξετάσουμε και να βρούμε νέες μεθόδους χρηματοδοτήσεως για τις υποανάπτυξη χώρες. Η διαφοροποίηση είναι όλο και πιο σημαντική στις χώρες αυτές. Προ 50 ετών ήταν απλώς φτωχέ, ενώ τώρα δεν ε, ισχύει. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη ε, διαπιστώνεται σε αυτές τις χώρες και η ιδίω στις χώρες της Αφρικής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υποκινήσουμε αυτή την οικονομική αύξηση και να φροντίσουμε όλοι αυτοί οι πολίτες να έχουν δικαίωμα να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και οι γυναίκες, ε, ε, οι ομάδες, τα περιθωριακά στοιχεία να μπορούν μπορούν να ε, συμμετέχουν σε αυτή την ε, ανάπτυξη ενώ άλλοι εποφελούνται περισσότερο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από ό,τι άλλος. Ορισμένοι απορρίπτουν τις γυναίκες μόνο λόγω του φίλου τους και εμείς που διαχειριζόμαστε δημόσιους πόρους πρέπει να λάβουμε μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Λαπόρτ να μου απαντήσει και να μου πει πώς ε, ε, θα μπορέσει κανείς να επιτύχει μία οικονομική ενσωμάτωση με διαφοροποίηση διότι οι δημόσιοι πόροι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη θα προέχει στις υποανάπτυξη χωρών, χώρες και γι' αυτό ε, εξετάζω το θέμα της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά τρόπον ώστε οι ε, τράπεζες αυτές να μπορέσουν ε, να συμβάλλουν εις την ενσωμάτωση των πολιτών και να τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή. Το 2012-2013 θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θα ήθελα Χάιτ να μου πει τι θα κάνει επί του θέματος αυτού. Δίνω τον λόγο στον κύριο Κάσμαν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχοντας ακούσει τους συναδέλφους, ε, θα ήθελα να κάνω μερικές σύντομες ε, παρατηρήσεις και θα σας αποδείξω ότι το να είσαι σύντομος είναι επί και Φυσικά και πρέπει να επιτυχούμε το 0,7 και πρέπει να αναφερθούμε σε αυτές τις χώρες. Αν θυμάμαι καλά αυτή, έχει εγκρίνει να υπάρχει μια ετήσια έκθεση όπου να αναφέρονται οι χώρες οι οποίες επέτυχαν ή δεν επέτυχαν το 0,7 του ΑΕ. Μια άλλη πρόταση εκτός από το φόρο των ε, χρηματικών συναλλαγών ήταν η πρόταση που είχα κάνει εγώ πολλές φορές ήταν ο φόρος ε, εμπορίας αγαθών όπως βαμβάκι, χαλκός, σιτάρι. Τα κέρδη από αυτό το εμπόριο θα πρέπει να επιστραφούν στα κράτη παραγωγής. Θα αποτελεί αυτό μηχανισμό, μηχανισμό παραγωγή, ε, ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πληρώνονται όμως φόροι σε αυτές τις χώρες από τις πολυεθνικές που υποστήριζουν αυτή την ανάπτυξη. Εμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι λοιποί θεσμοί μπορούμε να κάνουμε πολλά για να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και να είμαστε βέβαιοι ότι η ανάπτυξη ωφελεί αυτέ τι χώρε συζητώντας με τους φορολογικούς παράγοντες και να είμαστε βέβαιοι ότι οι αναπτυγμένες χώρες που ε, δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, πληρώνουν φόρους εκεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Πιστεύω ότι ήμουν αρκετά σύντομος, ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Tout à fait. Je vais encore passer. Συμφωνώ απολύτως. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Κορτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα-πρώτα κάτι θα πρέπει να διαπιστώσουμε όσον αφορά την πολιτική βούληση για αυτό το οποίο θα πρέπει ε, να πούμε σχεδόν στην κοινωνία ότι αυτό για το στόχο του 2015 είναι αυτό το 0,7% του ΑΕΠ, όμως θα πρέπει να, να, να πούμε ότι ε, αυτό είναι ο κοινό στόχο, 0,7-2015. Αυτό έχει σχέση με του στόχου τη χιλιετία, γιατί ακριβώ γνωρίζουμε ότι οι στόχοι ε, θα πρέπει να επιτευχθούν. Και επομένω αυτό ε, δείχνει το ότι ε, έχουμε ε, την, την, την, την, την, αποφασιστικότητα να βοηθήσουμε τι συγκρίσει τη στόχης και ότι θα το πετύχουμε με το 0,7. Θα πρέπει να μείνουμε στο 0,7 ούτως ώστε να μπορέσουμε έτσι να πετυχούμε τους μέλλοντες στόχους της ε, χιλιετίας. Είναι αυτό το θέμα μας, το, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει. Επίσης τώρα έχουμε μια σύντομη σκέψη ότι δηλαδή με την επίσημη στάση και αρρωγή της αμπτυξιακής βοήθειας μπορεί να μην ε, ε, λύσει το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως θα πρέπει να εντηρούμε τι προσθέσεις μα, Κύριε Λαγκάρπα, ε, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και από αυτό το κοινοβουλίο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες μεθόδους, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε κάποιες συμφωνίες, τόσο ώστε να γίνουν επενδύσεις, έργα, προγράμματα ε, να πετύχουν δική τη σωστή διακυβέρνηση και αυτό να γίνει στοχευμένα, ανατομέα. Γεωγραφική στόχευση επίσης. Αυτό νομίζω θα πρέπει να μας απασχολεί στο μέλλον όσον αφορά την αντιξιακή συνεργασία. Δίνω τώρα το λόγο ε, στην CDPM για τις απαντήσεις. Ποιος ξεκινάει η Κομισιόν. Σας. Ε, μας απευθύναν κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω σε αυτές για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση του κυρίου Κασμέ που αφορούσε την επιρροή που έχουμε στην αναβάθμιση των όντα στην Αφρική των επίσημων αναπτυξιακών αρρωγών. Αυτό αποτελεί απόφαση του κάθε κράτους μέλους του αν θα διαθέσει τα χρήματά του για όντα ή για, στρατιωτικές, ε, για θέματα ή για στέγαση. Δεν το επηρεάζουμε εμείς αυτό, ούτε τις περιοχές τις οποίες τα χρήματα θα δοθούν. Μπορούμε να κάνουμε προτάσεις αργότερα φέτος για το μέλλον της νέας αναπτυξιακής πολιτικής. Σίγουρα θα προτείνουμε κάποια διαφοροποίηση. Έχετε ήδη δει τις ε, προτάσεις του στο δημοσιονομικού πλαισίου για μετά το 2014 όπου ζητάμε εξέλιξη του EDF, το οποίο εστιάζεται στην Αφρική. Αυτά είναι όμως προτάσεις της Κομισιόν. Ε, τα περισσότερα πόσα μπορούμε να κάνουμε στην Αφρική ελέγχονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και από τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, στη συνέχεια κάνατε μια ερώτηση για το πώς μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση ε, σε χώρες όπως η Πολωνία και η Λετωνία. Η Κομισιόν ένιωσε πολύ άσχημα όταν τους έδειξαμε τα πρώτα γραφήματα και είδαν που βρίσκονται οι χώρες τους. Αυτό, ωστόσο, είναι το ίδιο με την πρώτη απάντηση. Οι χώρες αυτές έχουν την ευθύνη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έλαβαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στις 12 χώρες που εντάχθηκαν μετά το 2004 λένε ότι δεσμεύτηκαν για να προσπαθήσουν να επιτύχουν κάποια πράγματα. Δεν δεσμεύτηκαν για να επιτύχουν. Έτσι ισχυρίζονται. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία. Αυτή ήταν μια γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι 15 ε, παλιότερα μέχρι το 2002 Κατά την απόψή μου έχουμε πολλά να κάνουμε στη συνεργασία μας με τις κυβερνήσεις για να ε, κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η αναπτυξιακή συνεργασία. Δεν πρόκειται μόνο για πράξη αλληλεγγύης, αλλά για αντιμετώπιση των βασικών αιτιών ε, και όχι για να στηρίζουμε αυτές τις βασικές αιτίες, οι οποίες μετατρέπονται μετά σε μεταναστευτικές ροές και έχουν τεράστιες επιδράσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εργαστούμε πολύ για την ευαισθητοποίηση επειδή οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν ε, λιγότερη παράδοση ας πούμε στην αναπτυξιακή συνεργασία από τις υπόλοιπες. Ε, για τον κύριο Γκέρενς, ε, πολιτική βούληση. Έχετε απολύτως δίκιο. Ήθελα να προσθέσω επίσης η Φιλανδία επίσης πέτυχε το στόχο του 2010 και θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι και η Γαλλία σχεδόν τον πέτυχε. Ε, πρέπει να κάνει ακόμη ορισμένα πράγματα για να τον επιτύχει. Και εγώ εκπλήσωμαι όπως εσείς για τη Γερμανία. Ε, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στον Bundestag, υπάρχει κάποια διαρκής ε, πρωτοβουλία, κάποιο είδους ε, αναφορά εντός του Κοινοβουλίου, ώστε να ληφθεί υποστήριξη για το στόχο του 0,7%. Αυτό θα μπορούσε να σας δώσει μερικές ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε στα δικά σας εθνικά κοινοβούλια είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε παρόμοιε προσεγγίσεις και πρωτοβουλίε σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια για να ενισχύσουμε εντό των κοινοβουλίων την υποστήριξη προ του στόχου 0,7 ως ένα στόχο που θα επιτευχθεί πραγματικά και όχι απλώς για να γίνει μια προσπάθεια όσον αφορά την επερχόμενη έκθεση του EPCD ε, βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη για αύριο και δεν μπορώ να σας πω ε, σίγουρα αν ε, επικεντρώνομαστε προβολικά, στα βιοκαύσιμα στη γεωργία επειδή δεν είναι ο τομέας μου αλλά η έκθεση PCD θα ε, κυκλοφορήσει όσον αφορά την υπευθυνότητα θα υπάρχει και στην ατζέντα του Πουσάν και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία Αύριο θα μπορείτε με έναν ε, συνάδελφο αύριο να συζητήσετε, ε, συζητώντας για την προετοιμασία για το Πουσάν. Επίσης ρωτήσατε πως σκοπεύουμε να προβάλλουμε περισσότερο την εκθεσή μας στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Πολύ καλή ερώτηση, πρέπει να το εξετάσουμε. Έχουμε προσπαθήσει να προβληθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε γίνει πιο διαφανείς, έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια φέτος. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν περιλαμβάνεται ε, στην ατζέντα ε, για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, των ημερών Ευρωπαϊ... ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πάμε την εκθέση εκεί. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί με την ε, νεοσυσταθήσα ομάδα επικοινωνίας μας και μέσω των ε, ε, αντιπροσωπιών ε, και με τους ενδιαφερόμενους και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η επόμενη ερώτηση για το φόρο των οικονομικών συναλλαγών. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη είχαμε σκεφτεί ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις καινοτόμες πηγές που θα προσφέρει πολλά χρήματα σε σχέση με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες, αλλά βλέπω ότι στη δική μας την πρόταση της Κομισιόν για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ε, γίνεται πρόταση χρηματοδότησης του όλου προϋπολογισμού. Δεν γνωρίζω αν εντός της Κομισιόν θα υπάρξει όθηση για να εστιαστούμε στην κινητοποίηση αυτών των χρημάτων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ή για τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης των κλιματικών λαγών ή κάτι που να σχετίζεται με την ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν θα είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτό ποτέ θα υλοποιηθεί. Ε, δυστυχώς πολλά κράτη-μέλη έχουν ενδιασμούς όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Για τον κύριο Κάσμαν ήθελα να πω ότι ναι, υπάρχουν ε, και άλλες σημαντικές καινοτόμες πηγές που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε εκτός από όσα είπατε ο φόρος εμπορίας αγαθών και ο φόρος ε, εμπορίας ε, εκπομπών. Μόνο δύο κράτη-μέλη έχουν δώσει κονδύλια για χρηματοδότηση τέτοια σε αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε, αλλά και πάλι εδώ πρόκειται για απόφαση των κρατών μέλων. Μου άρεσε πολύ η ιδέα που προτείνατε να εκπονεί η Επιτροπή μία έκθεση κάθε χρόνο που θα αναφέρουμε τις χώρες που επιτυγχάνουν τους στόχους. Θα ήταν πολύ καλό θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μια έκθεση και από αυτή την πλευρά εδώ των ευρωπαϊκών θεσμών, γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο ακροατήριο, οπότε θα επικροτώ ιδιαίτερα αυτή την ιδέα. Ναι, στον Κορτές, ε, μιλήσατε για τα Εθνικά Κοινοβούλια, ήδη έκανα ένα σχόλιο για αυτό. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό αν μπορείτε να κινητοποιήσετε, να ευαισθητοποιήσετε τον πληθυσμό σε εσά ε, για τα όντα, για, την αίτια ε, για τις επίσημες αναπτυξιακές Αυτό που βλέπω λοιπόν από αυτή τη συζήτηση συζητήσαμε πολύ εδώ και το περισσότερο τα περισσότερα που είπαμε να αφορούσαν τα όντα. Ο κύριος Λαπόρτ. Ναι κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής. ίσως κάποιος δεν με κατανόησε καλά, ίσως ήμουν λίγο προκλητικός, είχα 8 λεπτό και έπρεπε να περάσω κάποιο μήνυμα. Φυσικά ε, οι επίσημες αναπτυξιακές αρρωγές, ODA, αποτελούν σημαντικό καταλήτη για την ανάπτυξη. Φυσικά θα πρέπει να προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους ε, που έχουμε θέσει έως το 2015. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το μήνυμα. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ενώ πρέπει να πετύχουμε αυτό το στόχο του 0,7% δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες πέραν των ODA η, από τη συζήτηση αυτή απορρέει ότι τίνουμε να επικεντρωνόμαστε συνεχώς στα ODA ενώ μπορούμε να ανακαλύψουμε και πολλά περισσότερα. Αισθάνομαι ότι η έκθεση υπευθυνότητα ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Αναφέρει όλες τις πιθανές ε, εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να μην εστιαζόμαστε υπερβολικά ή αποκλειστικά στη ODA και να δούμε πώς μπορούμε να κοινοτοποιήσουμε τους άλλους πόρους αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει καλύτερες επιδόσεις, να επενδύει περισσότερα αξιοποιώντας τις εναλλακτικές αυτές ε, ευκαιρίες χρηματοδότησης. Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο μεγέθη, Μερικέ φορέ έχουμε την τάση να μιλάμε μόνο για μεγέθη, για ποσά, αλλά αφορά και υπευθυνότητα. Εν τέλει, οι πολίτες και οι αναπτυσσόμενες χώρες θέλουν ε, οι δικές τους κυβερνήσεις να είναι υπεύθυνε και όχι οι δωρητές. Υπάρχει λοιπόν μια απευθεία σύνδεση. Αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε μεταξύ πολιτών, αναπτυσσόμενων χωρών και των κυβερνήσεών τους και το πώς αυτό μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω φορολογικών συστημάτων και άλλων εσωτερικών εγχωρίων μέσων που οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι πολίτες των αναπτυσσόμενων χωρών θα μπορούσαν να βοηθήσουν για την υπευθυνότητα των χωρών τους. Δεν είναι λοιπόν μόνο ευρωπαϊκή επιθυμία το να επενδυθούν περισσότερες προσπάθειες στις ίδιες αναπτυσσόμενες χώρες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό έχει και την υποστήριξη των θεσμών των αναπτυσσόμενων χωρών, επειδή η φυσιολογική αντίδραση που θα είχαν οι περισσότεροι από εμάς θα ήταν η Ευρώπη δεν θα πετύχει τους στόχους της, οπότε θα ρίξει τις ευθύνες στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη δική τους ανάπτυξη. Όχι, εν τέλει οι ίδιες οι αναπτυσσόμενες χώρες μέσω των δικών τους θεσμών έχουν δηλώσει με σαφήνεια ότι αποτελεί δική τους ευθύνη να προχωρήσουν ε, όσον αφορά αυτούς, αυτές τις πηγέ, πηγές, αναπτυξιακές πηγές ε, θα ήθελα να αναφέρω το συμβιβασμό της Τίνιδας. Ε, πρόκειται για ένα συμβιβασμό που επιτεύχθηκε νομίζω πριν από έξι μήνες στην Τινησία, στην Τίνιδα, από όλους τους ε, Αφρικανούς παραγόντες ε, για την προετοιμάζοντας το Πουσάν. Μία από τις συστάσεις κλειδιά ήταν ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την εξάρτηση από την αρρωγή. Ενώ αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η αρρωγή προς τις αφρικανικές χώρες, ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την εξάρτηση. Πρέπει να βρούμε ένα δρόμο ώστε να απεξαρτηθούμε αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το διεθνές εμπόριο και η επένδυση. Θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειες ε, ε, για κινητοποίηση των εγχώριων εσόδων που αντιστοιχούσαν το 2008 το δεκαπλάσιο της αρρωγής που έρε εντός της Επίρου. Για αυτό τον λόγο η Αφρική χρειάζεται δίκαια και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν για αυτό το πρόγραμμα και να επινοήσουν ε, επενδύσεις που θα βοηθήσουν ε, στην ανάπτυξη αυτό απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία επίσης των δωρετών ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικότερο δωρετή να προσπαθήσουν να υποστηρίξει αυτές τις χώρες ώστε να επαναπρογραμματίσουν την αρρωγή προς όφελος των τοπικών θεσμών που θα δημιουργήσουν πηγές αναπτυξιακής χρηματοδότησης μέσα στις εκάστοτε χώρες. Οι συζητήσει έτσι λοιπόν γίνονται πολύ πιο ενδιαφέρουσε ε, ε, και ειδικότερα οι ζωντανέ συζητήσει. Πέραν των ODA υπάρχουν τόσε πολλέ ευκαιρίε που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Οι φόροι οικονομικών συναλλαγών, συζητήθηκε ο φόρο ε, συναλλαγή εκπομπών, των φορεί επί αεροπορικών εισιτηρίων. Υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα από πηγές αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων. Α προσπαθήσουμε να τις εκμεταλλευτούμε προς όφελος του αναπτυσσόμενου κόσμου γενικότερα και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει περισσότερο σε αυτές τις εναλλακτικέ χρηματοδοτικές πηγές στο μέλλον επειδή έχουν περιγραφεί και τεκμηριωθεί με σαφήνεια σε αυτή την έκθεση accountability υπευθυνότητα. Α προσπαθήσουμε λοιπόν να τις υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όντως έχουμε, ε, ευχαριστώ, όντως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας Ξεκινάμε όμως τον προπολογισμό 2012. Έχουμε ήδη υιοθετήσει μία εντολή για τον τριμερή διάλογο με εισηγητή τον κύριο Γκέρενς. Έχουμε υποβάλει ορισμένες τροπολογίες στην Επιτροπή Προπολογισμού για τους πρώτους αριθμούς που έχουν μεταβιβαστεί από το Συμβούλιο. Αύριο τελειώνει η προθεσμία για τις τροπολογίες σχετικά με τον προπολογισμό αύριο Τετάρτη στις 17 και 30. Θα ψηφίσουμε στις 29 Αυγούστου και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι την κατάλληλη στιγμή σχετικά με ε, την, ε, το θέμα αυτό και συμφωνώ με τον κύριο Λαπόρτ. Πρέπει όμως να σας πω ότι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και η στάση της, του Συμβουλίου είναι ατυχής και επιμένω ότι είναι ατυχής διότι συνέχεια μας λέγουν ότι πρέπει να επιτύχουμε το 0,7% και πρέπει να υπάρξουν επίπεδα κλιμακοτά... και κάθε χρόνο πρέπει να αυξάνουμε το ποσό που θα διαθέτουμε για την ανάπτυξη και δεν καταφέρνουμε να καλύψουμε τους στόχους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να καλύψει τις δημοσιονομικές προοπτικές μέχρι το 2013 και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι ανακοινώσεις για το 2013 μέχρι 2020 που δεν είναι πιο ενθαρρυντικές από ό,τι έχουμε δει. Γι' αυτό κατ' εμέ υπάρχει ένα λάθος ως προς την ε, κατάρτιση του προγράμματος. Γιατί αν θέλουμε από τη μία πλευρά να πετύχουμε το 0,7 και από την άλλη πλευρά ε, διατυπώνουμε στόχους δημοσιονομικούς οι οποίοι εμποδίζουν και φρενάρουν αυτή την ανάπτυξη. Ε, είμαστε λοιπόν ε, ε, δεσμευμένοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο μας λέγει ότι δεν μπορεί να υπερβεί το 0,7% και πρέπει να υπάρξουν πολιτικές επιλογές και για το 2012 αυτό γίνεται κατά βάθος της αναπτυξιακή συνεργασία, συνεργασίας. Είναι δηλαδή το αντίθετο ακριβώς από αυτό το οποίο διακηρύσουμε και το έχει ε, δηλώσει, το είχα δηλώσει την ε, ε, πρώτη μου, στην πρώτη μου πολιτική παρέμβαση είπαμε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο το πρόγραμμα και η Επιτροπή μας απάντησε ε, καλά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είμαστε αρκετά απαιτητικοί και θέλουμε απλώς να αποκαταστήσουμε την κατάσταση στο επίπεδο που ήταν προηγουμένως. Γιατί λοιπόν να μειώσουμε το προϋπολογισμό των DCI. Ε, δεν βλέπω καμία πολιτική αιτιολογία για να μειώσουμε ε, σε αυτό το επίπεδο ε, και οι τροπολογίες μου αποβλέπουν στο να επανέλθουμε στον προϋπολογισμό, στο επίπεδο του προϋπολογισμού του 2011. Επίσης η Επιτροπή προτείνει ε, ε, ε, μία μεταφορά που θα ακουστήσει στο DCI 51 εκατομμύρια για το 2011. Έχουμε απευθύνει μία επιστολή στον πρόεδρο Λαμασούρ και η Επιτροπή επιπλέον και αυτό είναι ακόμη χειρότερο και συμφωνεί με αυτά που είπα στην αρχή να μειώσουμε κατά 100 εκατομμύρια τα DCI για το 2013. Είναι απαράδεκτο. Όσον αφορά την ε, συνεργασία με τις χώρες Λατινικής Αμερικής, Ασίας και Κεντρικής Ασίας, ε, εγώ ζητώ να αποκατασταθεί ο προπολογισμό. Δεύτερον, για την Παλαιστίνη που η Επιτροπή ζητά να μειώσουμε από 300 στα 200 εκατομμύρια και επιμένω να διατηρήσουμε το επίπεδο του 2011. Επίσης, ζητά να μειώσουμε από 65 σε 50 ε, εκατομμύρια και εγώ ζητώ για το AIDS να, ε, ε, και την φυματίωση να παραμείνουμε στα επίπεδα του 2011. Παντού λοιπόν είτε πιλωτικά προγράμματα είναι είτε άλλα ζητώ να διατηρηθούμε στα επίπεδα του προϋπολογισμού του 2011. Διότι αν θυμάμαι καλά η Επιτροπή είχε ζητήσει μία μείωση ενός εκατομμυρίου όσον αφορά τη σεξουαλική βία και τη βοήθεια στα θύματά της. Ε, ζητάει η Επιτροπή να ε, υπάρξει μία πίστοση 2,7 εκατομμυρίων υπέρ μίας προκαταρτικής δράσεως που είχαν προτείνει και οι συντονιστές και ε, ε, για τα υπόλοιπα θέματα η υγεία ε, να επανέλθουμε στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, τη διατήρηση του επίπεδου του 2011, ε, επισητιστική βοήθεια. Δεν νομίζω ότι η απειλή για την ε, επισητιστική ασφάλεια έχει μειωθεί και πρέπει να αποκαταστήσουμε τα αρχικά ποσά. Ανθρωπιστική βοήθεια, η Επιτροπή ε, θέλει να μειώσει, ενώ υπάρχει μία αυξημένη συχνότητα πιθανότητα καταστροφών. Ε, για την ασφάλεια μας ζητά να μειώσουμε τα 22 εκατομμύρια και ζητώ αποκατάσταση. Και τέλος, ε, ε, με συγχωρείτε, όπου σας είπα η Επιτροπή μέχρι τώρα διορθώνει ο κύριος Γιώρενς, πρέπει να μιλάμε για το Συμβούλιο. Όχι ότι είναι αμεμπτή η Επιτροπή, αλλά το Συμβούλιο είναι ε, αυτό που μας δημιουργεί τα προβλήματα. Όσον αφορά τώρα τις ε, διοικητικές δαπάνες, όλες οι αξιολογήσεις μας αποδεικνύουν ότι χρειάζεται ένα επίπεδο πόρων το οποίο ε, ανθρωπίνων πόρων, διότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ανθρώπινοι πόροι, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί η δράση και ε, διαφορετικά υπάρχει ε, μια ένα αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα. Ζητώ λοιπόν να μπορέσουμε να καταρτήσουμε αποτελεσματικά την ε, βοήθεια ιδίως όσον αφορά το προσωπικό το οποίο διατίθεται. Ε, ε, ε, επί όλων αυτών των θεμάτων θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και σας υπενθυμίζω ότι η υποβολή τροπολογιών είναι για τις 13 Ιουλίου 17 και 30. δεν έχουν ε, δικαιολογίες ούτε οι, Γερμα... ούτε οι Γάλλοι γιατί ακόμη και η 14... 14η Ιουλίου θα είναι ε, μετά από το πέρας της προθεσμίας ε, ε, υποβολής τροπολογιών και είμαι φίλος των Γάλλων. Η πρόοδος λέγει συμφωνώ απολύτως με όλα όσα είπατε κυρία ε, Πρόεδρε. Ε, ο κύριος Μπέρμαν. Ε, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ε, ο Σαλ Γκέρενς προσπαθεί να αποκαταστήσει τον προϋπολογισμό στην προτεραία κατάστασή του, ιδίως όσον αφορά δε την Παλαιστίνη. Δεν βλέπω κανένα λόγο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να μειώσουμε κατά 1 τρίτον την βοήθεια ε, ε, από 300 σε 200 εκατομμύρια και θα ήθελα να ξέρω τι αιτιολόγηση μπορεί να μας δίνει το Συμβούλιο. Θα ήθελα εδώ να θέσω αυτό το ερώτημα στο Συμβούλιο που παρίσταται. Γιατί αυτή η σημαντική μείωση. Οι Παλαιστίνοι πνίγονται κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, οικονομικά υπάρχει τραγική φτώχεια που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και είναι υπεραπαραίτητη η ευρωπαϊκή βοήθεια όχι μόνο στη Γάζα αλλά και σε, άλλα, ε, ε, σε άλλες περιοχές και υπάρχουν εδάφη που ποτέ δεν έχουν ε, βιώσει πραγματικές πολιτικές, προοπτικές και δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς την ευρωπαϊκή βοήθεια. Στηρίζω λοιπόν τον κύριο Γκέρενς για να αποκαταστήσουμε τον προϋπολογισμό και πιστεύω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Με εκπλήσει και με ενοχλεί ιδιαιτέρως η περικοπή για τις ε, ε, αποστολές παρακολουθήσεως των εκλογών γιατί αφελώς νόμιζα ότι όπου μπορεί να έχει ισχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ακριβώς στην στήριξη των ε, κρατών δικαίου που βοηθούν την δημοκρατία και ιδίω στην γένεσή της και αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων ένας τρόπος είναι η αποστολή ε, παρατηρητών ε, των εκλογών και δεν αντιλαμβάνουμε γιατί το Συμβούλιο αποφασίζει να περικόψει αυτό το ποσόν το οποίο θέλει να περικόψει κατά 5 εκατομμύρια που είναι το κόστος μίας αποστολής. Λοιπόν, ε, εάν δεν θέλουμε να στηρίξουμε τις ε, δημοκρατίες, ας το διακηρύξουμε εφταρσώς σχετικά με ε, την, ε, τα θέματα που ανέφερα θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλια του εισηγητή και του Συμβουλίου. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκέρενς για τη δουλειά του, για τις τροπολογίες για τις οποίες θα μιλήσω και σε λίγο επίσης. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερος για το πόσο με βοήθησε όσον αφορά την πρόταση για το πιλωτικό πρόγραμμα όσον αφορά την μητρική θνησιμότητα όσον αφορά συγκεκριμένα τις αφρικανικές εκείνες χώρες. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την αξιολόγηση, την εκτίμηση που έκανε για το πρόγραμμα των, που θα καλύψει τις χώρες εκείνες, για την πάνω στην βοήθεια. Θα επανέλθω όμως, πρέπει να του ευχαριστήσω. Ήταν στενή η συνεργασία και δεδομένη υποστήριξή του. Τσάλς, η προσέγγιση σου είναι 100% σωστή, με τίποτε. Δεν θα πρέπει να πέσουν θύματα της σε αυτέ οι χώρε. Σε σχέση με όσα γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην γειτονιά μας, οι ζωές των ανθρώπων στον επισόμενο κόσμο χρειάζονται τώρα περισσότερη προσοχή από ό,τι πριν την κρίση. Άρα είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έτσι τα θέματα αυτών των περικοπών και της απειλούμενης αναστολής εκτελέσεις των υπεσχεμένων και τα είπαμε και την περσμένη εβδομάδα, την Πέμπτη, για τις ε, μαζικές, τους μαζικούς ε, βιασμούς στο Κονγκό. Προσοχή, γιατί αν δεν κάνουμε κάτι θα είναι σαν ηθική χρεοκοπία. Άρα θα πρέπει τα θύματα αυτών των βιασμών να τα καλύψουμε υγειονομικά. Οπότε σωστό είναι να αυτά τα οποία λέμε να τα ακολουθούν συγκεκριμένες κινήσεις. Συμφωνώ για τόσα είπες όσον αφορά τις, ε, τους φορείς της ε, υγείας του διεθνής, για αυτό το ταμείο, για AIDS, ελονοσία, θυματίωση. Ε, πάει και πάλι συγχαρητήρια. Η πρόεδρος. Καλώς. Ναι, ναι, εκπληκτικά. Και τώρα το λόγο έχει πάλι και, και Όχι, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Αλλά η πράσινη σύμφωνη με το όσο είπατε 100% σύμφωνα με την έκθεση, συμφωνούμε με τις τροπολογίες Και επίση και ο σκιώδη ηγητή μα ο οποίο δεν μπορούσε να παραστεί, μου είπε να σας διαβάσω. Ευχαριστούμε. Κάσουμε ρέκα. Και εσύ και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρεν για τις τροπολογίε. Είναι αξιόλογε. Είναι αναγκαίε. Όσον αφορά τώρα την ενίσχυση προς την Παλαιστίνη. Υπάρχει εδώ κάποια ανακρίβεια. Στην δεύτερη φράση. Εκεί που έχουμε την θεολογική έκθεση. Βεβαίως και δεν πρέπει να συρρυκνώσουμε τα ποσά της ενίσχυσης, όμως εκεί στη δεύτερη φράση αναφέρεται ότι δεν πρέπει να μειωθεί. Όμως, έχουμε την τροπολογία που προβλέπει αύξηση της περσινής προοικοδότησης. Άρα, δεν ζητούμε τη σταθεροποίηση, τη διατήρηση, τη συνέχιση, ζητούμε την αύξηση της ενισχύσης τώρα όσον αφορά το Κονγκό. Τα συζητήσαμε στα κατεπήγοντα. Όσον αφορά δυστυχώς αυτούς τους βιασμούς, μιλάμε για 15.000 Πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό σε σχέση με πόσο γίνονται στο, στον κόσμο. Οι Κογκολέζοι δεν μπορούν να καλύψουν τα θύματα. Και όσον αυτά τα 2 εκατομμύρια δεν είναι και τόσο πολλά με δεδομένο το κόστος της αποστολής. Άρα θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι όπου έχουμε μπορέσει να βοηθήσουμε στο να γίνουν κάποιες ε, δημοκρατικές εκλογές, όπως εκεί. η αποστολή μας. Είναι λογικό να είναι ακριβή, είναι μακριά, δύσκολο να διοργανωθεί. Ε, και εάν θέλετε να συρρυκνώσουμε ή να καταργήσουμε την προσοχή σε κάποιες χώρες, ε, ναι, αν είναι για λόγους πολιτικούς, αλλά για λόγους οικονομικούς. Και φυσικά οπωσδήποτε πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα των βιασμών. Και τώρα ο κύριο Γκέρεν, ε, τελευταίος. Α, όχι, συγγνώμη, συμπαθώ Πρώτα η Κομισιόν. Σημειώνω. Είναι ο κύριος ε, Βοτρό για την ε, Γενική Διευθύνση των Προπολογισμών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ο Ζωακ Βαντρών από τη Γενική Διευθύνση Προπολογισμού η αρμόδια για τις εξωτερικές υποθέσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις παρατηρήσεις του. Δεν πρέπει να με την πρόταση της Κομισιόν και την ανάγνωση του Συμβουλίου. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εμείς ε, κάναμε μια πρόταση προϋπολογισμού που εντάσσεται σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που αποτελεί τον κανόνα του παιχνιδιού όπου ειδικά αυτό το πλαίσιο, αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να το υπερβούμε. Έχει παγιωθεί και αποφασιστεί από τις δύο δημοσιονομικές αρχές πριν από μερικά χρόνια. Αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σημαντικές δημοσιονομικές κρίσεις ε, σε όλα τα κράτη-μέλη μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σοφοί και αυστηροί και για τον κοινοτικό προπολογισμό και αυτό μας ε, επιβάλλεται ως κατάσταση συνεπώς οι προτάσεις μας λαμβάνοντας σε αυτό το πλαίσιο αλλά ε, και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα παρουσίασε ο εισηγητής. Επίσης υπάρχουν γεγονότα όσον αφορά την ε, αναπτυξιακή συνεργασία για τους διάφορους παγκόσμιους εταίρους που έχουμε. Επειδή η Κομισιόν, κυρία Πρόεδρε, ενδιαφέρεται ε, για την αναπτυξιακή ε, βοήθεια, αλλά υπάρχει και η βοήθεια προς τις υποψήφιες χώρες, προς τις τρίτες χώρες που ενδεχομένως δεν είναι αποδέκτες αναπτυξιακής αρρωγής. Η πραγματικότητα λοιπόν μεταβάλλεται συνεχώς από το 2006-2007 όπου ορίστηκε το πλαίσιο με κονδύλια αναφοράς που παρέμειναν ως είχαν και με περιθώρια τα οποία υπήρχαν και που η Κομισιόν κάθε, πρώτο, κάθε χρόνο προτείνει κατανομή ε, βάσει της ενότητας 4. Και υπάρχουν και κάποια μέσα ευελιξίας ε, είναι ε, το αποθεματικό επίγουσας βοήθειας που συχνά προτείνουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να αξιοποιήσουν για την αντιμετώπιση κρίσεων. Για παράδειγμα, θυμηθούμε την ΑΕΤ πέρυσι, όπου ε, κάναμε μια αίτηση την οποία δεχθήκατε. Ένα συνεπώς δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά πολύ διαφορετική εξέλιξη στην πραγματικότητα, όπως ε, αναδεικνύεται από το σημείο που ανέφερε ο κύριος Γκόρενς ε, για την αλλαγή του πλαισίου ορισμένων χωρών, οι οποίες πλέον ε, δεν είναι χώρες αποδέκτες αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά που οι ίδιες γίνονται χώρες ε, προσφέρουν βοήθεια και η Κομισιόν εκεί έχει δίκιο. Έχουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού, έχουμε ένα διορθωτικό ε, υπόμνημα επίσης, ε, φανταζούμε ε, μια διορθωτική επιστολή. Αυτή η διορθωτική επιστολή είναι πολύ θαραλέα, δείχνει την υποστήριξη, μια συγκεκριμένη προσπάθεια υπέρ της Αραβικής Άνοιξης για αυτές τις νεοεμφανιζόμενες δημοκρατίες και όπου προτείνουμε να δοθούν χρήματα, 400 εκατομμύρια το 2012 για αυτή την περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο στόχο επίσημης αναπτυξιακής ε, αρρωγής ε, για την Κομισιόν και για τον προπολογισμό της. Αυτές οι χώρες ε, είναι αποδέκτες της αναπτυξιακής αρρωγής. Όταν λοιπόν τους δίνουμε 400 εκατομμύρια, στατιστικά Ξέρω ότι αυτό δεν είναι πάντα το πιο σημαντικό, αλλά ηθικά έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά ε, την αναπτυξιακή αρρωγή. Όσον αφορά αυτή τη διορθωτική επιστολή, θα ήθελα να επιμείνω στην ε, αλλαγή κατεύθυνση που προτείνουμε μέσα σε αυτή την επιστολή, δηλαδή ότι ορισμένες ε, χώρες και όσον αφορά Ε, το, αυτό το έμβασμα 20 που ανέφερε ο εισηγητής ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι χώρες για τις οποίες προτείνουμε να υλοποιηθεί η αρρωγή δεν είναι χώρες που ενδιαφέρονται για τη βοήθεια αυτή είτε χώρες που εξάγουν πετρέλαιο είτε χώρες για τις οποίες, ε, με τις οποίες έχουμε συνεργασία όσον αφορά εκπαιδευτικά για παράδειγμα θέματα και που συνεχίζεται αλλά και τα κρατημέλη συμμετέχουν σε αυτή την αρρώγη. Το Μεξικό λοιπόν, η Βραζιλία, η Βενεζουέλα μεταξύ άλλων, η Ινδία και η Ταϊλάνδη ε, προτείνουμε ε, η αρρωγή προς αυτές να ε, μεταβληθεί και να πάει προς τις χώρες της Νοτιού Μεσογείου μέσα σε, στους μήνες που ακολουθούν την ε, μείζωνα κρίση που έλαβε χώρα σε αυτό το μέρος του κόσμου. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγήτη που υποστήριξε την αποκατάσταση της ε, διοικητική στήριξης. Την έχουμε... Ε, η Κομισιόν υποστηρίζει αυτή τη διοικητική στήριξη έχουμε προτείνει μια περιορισμένη αύξηση του χαρτοφυλακίου που μας ε, ε, έχει ανατεθεί να διαχειριζόμαστε ε, στην έδρα μας αλλά και στις αντιπροσωπείες. Αυτά ήθελα να σας πω εν συντομία και ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την υποστήριξή σας, για την αποκατάσταση των κονδυλίων μας ε, σε σχέση με τα όσα προτείναμε στο σχέδιο προϋπολογισμού και στη διορθωτική επιστολή. Ευχαριστώ κύριε Βόντρε. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με όσα είπατε, αλλά θα δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο Μπέρμαν και μετά στον κύριο Γκέρνς, ο οποίος θα ολοκληρώσει. Ίσως δεν πρόσεξα καλά, αλλά δεν άκουσα απάντηση για το Παλαιστινιακό ζήτημα ξανα, ε, να σας ξαναδώσω το λόγο για ένα λεπτό. Ε, έχει δίκιο ο κύριος Μπέρμαν, ξέχασα να απαντήσω. Όντως ο όγκος τον οποίο προτείνουμε στο σχέδιο προπολογισμού ε, ανταποκρίνεται σε ένα υψηλότερο ποσοστό από αυτό το οποίο προβλέπεται στον πολιετή φάκελο ο οποίος ψηφίστηκε για την περίοδο 2011-2013 και που έγινε αποδεκτή από τα διάφορα θεσμικά όργανα ε, στα πλαίσια της δημοκρατικής αναθεώρησης των προγραμμάτων που ε, έχουν σημασία στρατηγικής ενισχύσεως της περιοχής λοιπόν, έχουμε από 300 εκατομμύρια όντως εμείς προτείνουμε περικοπή ε, κατά 1 τρίτον στα 200 εκατομμύρια διότι υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί εκ των οποίων μπορεί να επωφεληθεί η Παλαιστίνη. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα μίας γραμμής αλλά πολλαπλών δυνατοτήτων και θεωρούμε ότι η Παλαιστίνη πλέον εφόσον έχει ε, μία γραμμή ε, δημοσιονομικής επιβίωσης που προσφέρεται εις ε, την Παλαιστινιακή Αρχή θέλουμε να καταρτήσουμε στην Παλαιστίνη πραγματικά προγράμματα και όχι μόνο να καλύπτουμε τις ανάγκες του στο τέλος του μηνός. Για να γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξουν προγράμματα, ξεμπλοκάραμε ορισμένα δημοσιονομικά κεφάλαια τα οποία είχαν κατασχεθεί η ε, στο παρελθόν από τις Ισραηλινές αρχές και αυτό είναι σημαντικό και πολλές φορές ε, αυτό μπορεί να ε, αντιπροσωπεύει το ποσό το οποίο μας επιπλήτεται ότι μειώσαμε. Είναι ευκαιρία να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αντικαθιστά τους φυσιολογικούς πόρους της Παλαιστινιακής Αρχής η οποία πρέπει να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σαν κυβέρνηση η οποία λειτουργεί. Ε, ποτέ δεν είδα κάποιον να εκφραστεί και να μην, το να μην καταλαβαίνει γαλλικά αφού του μιλώ. Εφόσον μου λέτε ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες χρηματοδοτήσεως, που... ποιες είναι αυτές οι άλλες δυνατότητες και από πού καλύπτονται. Είναι ένα προπέτασμα καπνού. Ε, ε, πρόκειται για την πολιτική γυτνιάσεως που είναι ένα μέσο το οποίο ενισχύεται και για ε, τρία χρόνια προτείνουμε να υπάρξει μία χρηματοδότηση σε 1,4 δισεκατομμυρίων με ανακατατάξεις και ε, είναι πάλι ένα υψηλό ποσό το οποίο είναι υψηλότερο από την ε, πολιετή ε, πρόοδο που έχει προβλεφθεί για το 2011-2013. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να καλυφθεί από την πολιτική γυτνιάσεως αυτό το θέμα και δεν θέλουμε μόνο να υπάρχουν μεταφορές δημοσιονομικές απλώς για να βοηθήσουμε και να καλύψουμε την Παλαιστινική ε, ε, αρχή στην κανονική της λειτουργία. Το προπέτασμα καπνού δεν αναφέρεται μόνο στην Παλαιστίνη, ε, αναφέρεται σε ολόκληρη την Αραβική Άνοιξη. Η Παλαιστίνη συμμετέχει εις την στην πολιτική γυτνιάσεως και σαν την, την Ισία και τις άλλες χώρες θα μπορέσει να υποφεληθεί των ενισχυμένων φακέλων που προσφέρουμε. Ο κύριος Γκέρενς σχετικά με το προπέτασμα καπνού, εγώ θα ήθελα να πω ότι παραμένει ομιχλώδης η κατάσταση διότι ε, δεν νομίζω ότι έχουμε ικανοποιηθεί αλλά υπάρχει κάποια ε, διαφωνία και δεν συνεννοούμαστε. Ε, μου φαίνεται πιθανόν αυτό το οποίο μου λέτε αλλά εγώ είχα ζητήσει να γνωρίσω τι θα γίνει γιατί ενοχλήθηκα για τη μείωση καταρχήν. Αλλά θα επανασυνδεθώ με τους υπευθύνους και να δω εάν μπορούν να με καλύψουν. Ε, δεν αμφισβητώ την καλή σας πίστη, αλλά θέλω να το ακούσω από τον υπεύθυνο. Δεύτερον, όσον αφορά την επιτόπου κατάσταση, όντως υπάρχουν χώρες οι οποίες σήμερα είναι υπό ανάπτυξη, αλλά δεν είναι ίσως αναδυόμενος, έχουν αναδυθεί ήδη. Άρα η συζήτηση η οποία γίνεται εδώ δεν, ε, είναι, ε, ε, δεν μας βοηθάει διότι μιλάμε για ενίσχυση των αναδειωμένων χωρών, για βοήθεια των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και βλέπουμε ότι λιγότερο από τα ίμιση των κεφαλαίων ε, πρέπει να καλύπτουν χώρες ε, λιγότερο προηγμένες που χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση. Και αυτό δεν είναι κάτι που ίσως θα καλύψουμε τώρα στην παρούσα φάση της δημοσιονομικής συζητήσεως, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να ε, ξαναεξετάσουμε εκ του σύνεγγυς. Και όλα αυτά ε, δεν, ε, δεν καλύπτονται από τον όγκο ενισχύσεως. Πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει το 0,7% για να υπάρξει μία βαθμιαία ανάπτυξη μέχρι το 2015, διότι διαφορετικά δεν αποδίδουν τα δημοσιονομικά κεφάλαια και πρέπει η εξέλιξή μας να είναι ανωδική και όχι καθοδική. Ευχαριστώ την κυρία Κέλλερ για τη βοήθειά της και τον κύριο Κασμάρεκ και θα ήθελα να σας πω ότι ιδίως να πω ε, στον κύριο Κάσμαν ο οποίος με επένεσε τόσο πολύ ότι όταν είναι κανείς πολιτικός ηθήνων πάντοτε έχει φιλοδοξίες αλλά σε ευχαριστώ Μάικελ με ευχαρίστησε και με καθησυχάζει αυτό που μου είπες θέλω να έχω φιλοδοξίες και ε, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι για σοσιαλιστής ο κύριος Κάσμαν δεν είναι και κακός και η τελευταία μου παρατήρηση αναφέρεται εις ε, την περίεργη στάση της κυρίας Άστον, της Λέδης Άστον, διότι ποτέ δεν μιλά περί του ε, ε, προϋπολογισμού θέλει να ελέγξει την ε, πολιτική αναπτυξιακή συνεργασίας, κινητοποιεί ε, τους και συζητά με τους εθνικούς ε, υπευθύνους. Δεν είχαμε συναντήσει ούτε τον κύριο Μισελ όταν ήταν η Βελγική Προεδρία, ούτε τον υπεύθυνο της εξερχομένης Προεδρίας. Θα ήθελα λοιπόν τουλάχιστον η κυρία να μας εξηγήσει τη θέση της, διότι είναι αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετέχει στις υπηρεσίες που κατακρίνουμε και σαν υπεύθυνη ε, της εξωτερικής δράσης έχει δύο σωσίες όσον αφορά τη θέση την οποία λαμβάνει στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να μας εξηγήσει τη θέση της, γιατί έχει μία περίεργη ε, θέση η οποία αφήνει πολλά ερωτηματικά. Εφόσον λοιπόν είναι η πρώτη πολιτική υπεύθυνο, θα πρέπει αυτή να επικροτήσει και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Συνένεση θα αποτελεί απλώς ένα δόγμα δίπλα εις ε, τη διακήρυξη της Άκρα και άλλες. Είναι λοιπόν χρήσιμο για τη συζήτηση αυτό και για τις επόμενες ε, προθεσμίες που έχουμε μέχρι ε, τις ελεύσεις που προβλέπονται. Η κυρία Άστον λοιπόν μου λέγεται ότι θα έρθει σε μία επόμενη συνεδρίασή μας στο Φιδινόπορο. δεν έχω ακόμη την ημερομηνία, αλλά θα την ρωτήσουμε όταν θα έρθει εδώ. Νομίζω ότι είναι 12 και 20, λίγη η συνεδρίασή μας και θα, θα επανέλθουμε στις 3. Σας εύχομαι καλή όρεξη.